Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Μπορεί να μην έχουμε φως, έχουμε όμω μικρόφωνα. Έχουμε διερμηνία. Οπότε μπορούμε να αρχίσουμε. Και το φως θα έρθει αργότερα, ελπίζω. Δεν ξέρω γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, κηρύσω την έναρξη τη συνεδρίαση της επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης που θα είναι σήμερα και αύριο. Αρχίζουμε με την έγκριση τη ημερήσιας διάταξη. Σχόλια με τη ημερήσιας διατάξεως. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της κυρίας Νταμάτο, που πρέπει να λείψει για λίγο, γιατί ψηφίζει σε άλλη επιτροπή, θα θέλαμε να ζητήσουμε την αναβολή του 5 για μια μελλοντική συνάντηση σχετικά με το πολιετές δημοσιονομικό. Θεωρούμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ύψος της προχρηματοδότησης θα επηρεάσει πάρα πολύ τη σύνταξη της συμφωνίας. Δεν υπάρχει λοιπόν μια συμφωνία. Αν δεν υπάρξει συμφωνία για την μετακίνηση, ε, ζητάμε να ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία και όχι η έκτακτη την οποία προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you very much. I... Ευχαριστώ. Πρέπει να ενημερώσω τα μέλη της Ρέτζη ότι έχω λάβει μια επιστολή από την κυρία Νταμάτο εξέφρασε τις αντιρρήσεις της για το σημείο 5 της ημερησίας διατάξεως. Όταν φτάσουμε στο 5 είχα σκοπό να παρουσιάσω την επιστολή. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχουν τα πράγματα, εάν δεν υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις από πλευράς υπολείπων πολιτικών ομάδων, θα μπορούσα κάλλιστα να αποφασίσω την αναβολή του 5 και την διεξαγωγή ε, της ε, συζήτησης αυτής στους συντονιστές για να δούμε ακριβώς ε, πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον με το συγκεκριμένο ντοσιέ γιατί έχουμε την απόφαση των συντονιστών για τέτοιου είδους διαδικασίες. Αυτή είναι η εντολή την οποία έχουμε πάρει από τους συντονιστές και η εντολή αυτή μπορεί να αλλάξει αλλά μόνο από τους συντονιστές. Λοιπόν, τώρα επιτρέψτε μου να αφαιρέσω το σημείο 5 από την υπηρεσία διάταξη και να συμπεριλάβουμε αργότερα τη συζήτηση αυτή σε επίπεδο συντονιστών, αν συμφωνείτε. Ευχαριστώ πολύ. Με αυτή την αλλαγή λοιπόν διαγράφουμε το 5. Μπορούμε να υιοθετήσουμε την υπόλοιπη μερίσια διάταξη. Ευχαριστώ. εγκρίνουμε τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων της 27ης Σεπτεμβρίου του 2018. Ε, είναι διαθέσιμα online τα πρακτικά αυτά και αν δεν ε, ανακοινηθούν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θεωρούνται δεκτά. Ελπίζω να έχω ανακοινώσεις στην επόμενη συνάντηση, σε δέκα μέρες, στην επόμενη συνεδρίαση μάλλον. Και τώρα περνάμε αμέσως στο πρώτο θέμα της κανονικής ημερήσιας διάταξης, πρόταση γνωμοδότησης για την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Η κυρία Μάλετιτς είναι η συγγήτριά μας. Έχουμε και τους σκιώδεις παρόντες, νομίζω, βλέπω και άλλους. Έχετε κυρία Μάλετιτς τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που είμαι εισηγήτρια για ένα τέτοιο θέμα, ιδιαίτερα για τους νέους που δημιουργούν ευκαιρίες ε, δημιουργούνται ευκαιρίες για την απασχόλησή τους στα πλαίσια της εθελοντικής εργασίας. Στην γνωμοδότηση υπογραμμίζω ότι οι δραστηριότητες αλληλεγγύης δεν θα πρέπει να περιορίζονται στην κατάρτιση, την εκπαίδευση και την απλή απασχόληση, θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, επαρκούς ποιότητας μάλλον, και ε, κοινωνικά χρήσιμες. Αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι είναι σημαντικό με τον φάκελο αυτό να καταστήσουμε δυνατό στα πλαίσια της διαδικασίας εφαρμογής την λήψη των απαιτούμενων μέτρων. Γιατί έχει σημασία οι συμμετέχοντες στις ε, εθελοντικές αυτές δραστηριότητες να αποζημιώνονται σαν παράδειγμα να καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησής τους, να τους δίδεται pocket money, ένα είδος ε, χαρτζιλίκι. Υποστηρίζω επίσης ότι όποια μονάδα, ενότητα, σύλλογος θέλει να συμμετέχει στις δραστηριότητες αυτές, θα πρέπει να παίρνει και ένα σήμα ποιότητας στον τομέα της αλληλεγγύης. Και αυτό βέβαια θα πρέπει να ελέγχεται σε τακτική χρονική βάση. Νομίζω ότι η δημοσιοποίηση και διάδοση των ε, ευκαιριών και των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται να τονισθούν ακόμα περισσότερο, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Να γνωρίζει ο κόσμος πώς λειτουργεί το πρόγραμμα αυτό και τι αποδίδει. Και σε σχέση με την απλούστευση την οποία αναφέρθηκα, απαιτούνται περαιτέρω, απαιτείται περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών διαδικασιών έτσι ώστε να γίνονται σωστές επιλογές σε επίπεδο κόστους και να υπάρχει έτσι μεγαλύτερη άνεση για τους δικαιούχους. Επίσης καθορίζονται συγγνώμη, τα επίπεδα ελέγχου τα οποία θα πρέπει να γίνονται από τις εθνικές αρχές αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις απαιτήσεις απλούστευσης ή απλοποίησης και να μην επιβαρύνουμε το σύνολο των συμμετεχόντων. Σας ευχαριστώ κυρία Μάλετιτς. Θα δώσω το λόγο στους Κιώδης. Ο κύριος Χαουόργ δεν είναι εδώ. Ο κύριος Κοσόφσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι πεπισμένος ότι το σώμα αλληλεγγύης θα είναι μια καλή ευκαιρία για τους νέους να προχωρήσουν σε εθελοντική εργασία στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής οικονομίας. Θα τους δώσει την δυνατότητα να αναπτύξουν και δικά τους προγράμματα αλληλεγγύης να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ε, προσωπική τους ε, εξέλιξη και ανάπτυξη και θα βελτιώσει επίσης και τις δυνατότητες απασχόλησης. Θα στηρίξω λοιπόν την πρόταση για την περίοδο 21-27. Πρέπει να επενδύσουμε στους πολίτες της Ευρώπης και είμαι ικανοποιημένος γιατί προβλέπονται δράσεις για την βελτίωση των πολιτών στις κοινωνικές εξελίξεις. Ε, με ικανοποίηση επίσης βλέπω και τις ευκαιρίες οι οποίες δίδονται ε, στους νέους οι οποίοι δεν έχουν πάρα πολλές δυνατότητες και θα πρέπει να υπάρξουν ε, λύσεις εδώ έτσι ώστε να διευκολύνουμε την κοινωνική επανένταξη με τρόπο ε, ώστε οι κάτοικοι των λιγότερο ευνοημένων περιοχών να μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα αλληλεγγύης. Πρέπει να εντοπίσουμε σωστά λοιπόν τις κοινωνικές αυτές κατηγορίες των νέων και να τις ενεργοποιήσουμε. Όπως είπα θα αναπτύξουν τις ε, κοινωνικές τους ικανότητες σε πολλούς τομείς της κοινωνίας. πρέπει να στοχεύσουμε τους πολίτες που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, είναι λιγότερο ευνοημένοι σε κοινωνικό επίπεδο και θα πρέπει βέβαια να διαφοροποιήσουμε πλήρως την εθελοντική δραστηριότητα από την επαγγελματική δραστηριότητα. Δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες της εθελοντικής εργασίας σαν εναλλακτική δραστηριότητα σε περίπτωση που υπάρχουν ε, κενές θέσεις πλήρους απασχόλησης. Μπορούν να βοηθήσουν λοιπόν οι αλληλέγγυοι και στον τομέα της φροντίδας των ηλικιωμένων, της φροντίδας ε, των αναπήρων κτλ. Αουστρεβίτσιος, ο επόμενος κοιόδης, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μάλετιτς για την εξαιρετική της δουλειά στα πλαίσια της δημιουργίας του European Solidarity Corps. Εγώ υποστηρίζω πολλές από τις προτάσεις της παρουσίασης. Αυτό το οποίο ξεχωρίζει λίγο είναι η ιδέα ότι η ετικέτα αυτή ποιότητας αλληλεγγύης θα πρέπει να ανανεούται αναδιετία. Και αναφέρομαι εδώ στην τροπολογία 18. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει περιοδικά. Αυτό ίσως να μην είναι πολύ συγκεκριμένο, αλλά η διετία της ε, εισηγήτριας θα δημιουργήσει πολύ γραφειοκρατία θα γίνονται συνεχείς αξιολογήσεις ε, για τις συμμετέχουσες οργανώσεις. Εάν προσπαθήσουμε λοιπόν να βοηθήσουμε και τις τοπικές οργανώσεις, μικρές οργανώσεις να συμμετέχουν, θα πρέπει τα γραφειοκρατικά άχθη να χρησιμοποιούνται μεν, να υπάρχουν μεν, αλλά όχι ε, να είναι επιβαρυντικά. Συνεπώς λοιπόν υπάρχει κίνδυνος να απολεστεί η αρχική χρήσιμη ιδέα λόγω της ε, διοικητικής δυσκολίας και της περιπλοκότητας. Να ευχαριστήσω την κυρία Μάλετιτς λοιπόν για την πολύ καλή της εργασία. Νομίζω ότι θα βρούμε τελικά κάποιες ικανοποιητικέ λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος σκιώδης ε, είναι από πλευράς των πρασίνων, όχι δεν υπάρχει. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Η κυρία Αντινόλφη Νομίζω ότι το Σώμα Αλληλεγγύης είναι ένα σωστό πρόγραμμα, μια σωστή πρόταση και πρέπει να υποστηριχθεί διότι επιτρέπει να θέσουμε σε πράξη τις αξίες της Ένωσης. Αλλά θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες τις οποίες θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε με τις συγκεκριμένες τροπολογίες. Δεν είμαι πεπισμένη για την δυνατότητα χρηματοδότησης όχι μόνο εθελοντικών δραστηριοτήτων αλλά και εργασιακών ε, δραστηριοτήτων όπως τα στάζ και οι συνοπτικές χρονικά συμβάσεις. Αυτό ε, στρεβλώνει την έννοια της αλληλεγγύης και θα μπορούσε να δείξει ε, ότι θα ήταν λανθασμένο βέβαια, το πρόγραμμα αυτό αντιμετωπίζει και την ανεργία. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά τις χώρες της Νότιας Ευρώπης ε, και απαιτείται εδώ δραστηριοποίηση στους τομείς έβρεσης θέων απασχόλησης, θέσεων απασχόλησης. Θα πρέπει επίσης στα πλαίσια της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνονται συμβάσεις εργασίας δίμηνες. Αυτό είναι απαράδεκτο και εγώ θα ήθελα να μην υπάρχει καμία σχέση της πρότασης με θέματα εργασίας. Και επίσης ε, σε ποιο βαθμό θα μπορούσαν οι κερδοσκοπικές οργανώσεις να συμμετέχουν στα προγράμματα. Αυτό δημιουργεί κινδύνους κατάχρησης, εκμετάλλευσης των νέων από πλευράς του ιδιωτικού τομέα. Να χρησιμοποιούν τους νέους οι επιχειρήσεις δωρεάν μεγιστοποιούν τα κέρδη τους και είναι πλήρως άσχετοι με την ευγενή δραστηριότητα της εθελοντικής εργασίας. Δημιουργούνται παράδεκτες καταστάσεις, παράδοξες καταστάσεις και μια μεγάλη εταιρεία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους μέσα μόνο και μόνο για να υπογραμμίσει τον κοινωνικό της χαρακτήρα και να μην επηρεάσει όμως θετικά τα κοινωνικά προβλήματα. Σε σχέση με το πρόγραμμα 2018-2020 που προβλέπει μια ανακατανομή του προϋπαλογισμού ανάμεσα στο κομμάτι της απασχόλησης και στο κομμάτι του εθελοντικού 10% από τη μία, 90% από την άλλη στην πρόταση που γίνεται τώρα δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός σε δημοσιονομικό επίπεδο. Ελπίζω ότι πρόκειται για μια παράληψη και όχι για μια συγκεκριμένη και σκόπιμη πρόταση. Ανάμεσα στις δύο αυτές διαφορετικές κατηγορίες δημιουργούνται πιθανώς φαιές περιοχές μέσω των στάζ και των σύντομων συμβάσεων απασχόλησης. Μοναδικός στόχος του προγράμματος θα πρέπει να είναι η εθελοντική απασχόληση. Το πρόγραμμα θα πρέπει να εγγυηθεί την προσβασιμότητά του σε όλους όσους αντιμετωπίζουν handicaps και θα πρέπει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες συμμετοχής σε αυτού του είδους τις εμπειρίες και οι προερχόμενοι από λιγότερο ευνοημένες κοινωνικο-οικονομικά ομάδες και θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα απόσυρσης της ετικέτας ποιότητας όταν διαπιστώνονται καταχρήσεις. Η εθελοντική απασχόληση πρέπει να είναι ο μοναδικός στόχος του προγράμματος που θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε η αδίποτε μορφή σύγχυσης με την απασχόληση. Ευχαριστώ. Αυτές ήταν οι παρουσιάσεις των σκιωδών. ο Σκιώδης ε, των Σοσιαλδημοκρατών παρουσίασε τις απόψεις της ομάδας του στην κυρία Μάλετη, στην εισηγήτρια. Είναι ενήμερη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο μέλος το οποίο θα ήθελε να πάρει μέρος στη συζήτηση. Καλώς λοιπόν θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Αναστόπουλος. Ελπίζω να το είπα σωστά. Η κυρία Αναστοπούλου, ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή ευχαριστεί την εισηγητρία για το σχέδιο γνωμοδότησης. Εκτιμούμε τις προσπάθειές σας προκειμένου το σώμα αλληλεγγύης να λειτουργήσει καλύτερα με απλοποίηση. Και θέλουμε να πούμε ότι στην τωρινή υλοποίηση ήδη χρησιμοποιούμε την απλοποίηση χρησιμοποιούμε κατά αποκοπή ποσά, αποζημίωση βάση μονοδιαίου κόστους, οπότε έχουμε ήδη αρχίσει μια διαδικασία απλοποίησης που θα συνεχιστεί βέβαια και στο προσεχές πρόγραμμα. Και πάντα με το πνεύμα της απλοποίησης συμφωνούμε με τους ισχυώδεις εισηγητές που είπαν ότι διευκρινίζοντας ότι το σήμα ποιότητας πρέπει να αξιολογείται κάθε δύο χρόνια, αυτό μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον άχθος θα είναι πιο δύσκολο για τις εθνικές υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους γιατί ήδη παρακολουθούν τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται επί τόπου. Είμαστε βέβαια ανοιχτοί να συζητήσουμε μαζί σας παρετέρω τα ζητήματα όσο προχωρά καιρός. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μάλεβιτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις εισηγητές και περιμένω τις τροπολογίες τους. Σίγουρα θα καταλήξουμε σε καλό συμβιβασμό. Τονίζω όμως ότι πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό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

Είναι τέσσερις παρατέταρτο. Τώρα έχουμε και φως και ήχο. Έχουμε και τη στήριξη των διερμηνέων, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Σταματήσαμε όταν η κυρία Μαλέτιτς τελείωνε την παρέμβασή της μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του δικού της θέματος. Είχαν μιλήσει σκιώδης ε, εισηγητές, είχε μιλήσει εκπρόσωπο της Επιτροπής. Το μόνο που μένει να πω είναι ότι προτείνω η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών να είναι στις 12 το μεσημέρι την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου. 12 το μεσημέρι την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου. Τώρα, Συνεχίζουμε και περνάμε στο επόμενο θέμα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Είπαμε ότι αναβλήθηκε το σημείο 5 και θα συζητήσουμε στους συντονιστές τι θα κάνουμε με αυτό. Και περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι ο κατεξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την κατάρτιση του καταλόγου δικτών για την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 1082 του 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει το σχέδιο κατά εξουσιοδότηση κανονισμού με τον κατάλογο των δικτών και έχουμε τρεις μήνες στη διάθεσή μας που μπορεί να παραταθεί η περίοδος αυτή για άλλους τρεις μήνες σε περίπτωση που έχουμε ένσταση. Εάν δεν υπάρξει ένσταση, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τον ε, κατεξουσδότηση κανονισμό. Λοιπόν, η Επιτροπή πρώτα απ' όλα θα μας παρουσιάσει αυτή την πράξη και μετά θα παρέμβουν και οι ευρωβουλευτές για να σχολιάσουν ή να υποβάλουν ερωτήσεις. Παρακαλώ. Φαν Μπρέσκα. Εσείς είσαστε υπεύθυνο κύριε Φανμπρέσκα. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα. Θα κάνω μια πολύ σύντομη παρουσίαση. Όμως, επειδή πρόκειται για ένα τεχνικό εγχείρημα, θα ήθελα να πάμε λίγο πίσω και να μας υπενθυμίσω περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται λοιπόν για ένα νομικό εργαλείο που διευκολύνει τη διασυνοριακή συνεργασία. Δημιουργήθηκε πριν από 10 χρόνια περίπου και επιτρέπει στις περιφερειακές και τοπικές αρχές διαφορετικών χωρών μελών από κοινού να δημιουργήσουν ε, κάποια σώματα συνεργασίας ώστε να φέρουν σε πέρας κάποια προγράμματα, υπηρεσίες κλπ. Αυτό που ίσως εσείς να ακούσει ένα πρόγραμμα για διασυνοριακό νοσοκομείο που είναι στα σύνορα Ισπανίας και Γαλλίας. Και εκεί αντί να δημιουργηθούν δύο διαφορετικά νοσοκομεία, δημιουργήθηκε ένα, μία νοσοκομιακή μονάδα που εξυπηρετεί και τις δύο χώρες. Και τη διαχείριση το οποίο έχει ακριβώς ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας. Η Επιτροπή πρότεινε και τον ε, διασυνοριακό ε, μηχανισμό συνεργασίας που είναι κάτι διαφορετικό. Ε, αυτό που κάνει αυτό το δεύτερο είναι ότι επιτρέπει οι κανόνες που ισχύουν σε μία χώρα να ισχύσουν για συγκεκριμένα προγράμματα στην γείτονα χώρα, εφόσον είναι κοινού οικονομικού συμφέροντος. Τώρα, ο κανονισμό αυτό Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκού Δαφική Συνεργασία επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει κατεξοδότηση πράξη με κατάλογο δικτών προκειμένου να μπορέσει να αξιολογήσει τον ε, κανονισμό αυτό. Και αυτό ακριβώς είναι που έχετε και εσείς ε, μπροστά σας σήμερα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για την κατεξουδότηση αυτή πράξη. Απλώς θα σας πω ότι έχουμε πέντε διαφορετικές ομάδες δικτών που έχουν να κάνουν με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη βιωσιμότητα και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτούς τους δείκτες τους έχετε στο παράτημα. Το ερώτημα βέβαια είναι γιατί τους χρειαζόμαστε. Και η απλή απάντηση είναι ότι αποτελούν τη βάση προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει έκθεση, να εξετάσει δηλαδή την εφαρμογή στην πράξη του κανονισμού που εγκρίθηκε πριν από μερικές εβδομάδες και αποστάλλει και στο Κοινοβούλιο και να υπογραμμίσει κάποια συμπεράσματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια κλπ. Έχουν αυξηθεί χώρες που συμμετέχουν από 48 σε 72, κατά 30% δηλαδή από το 2014 μέχρι σήμερα. Πράγμα που δείχνει ότι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία τέτοιου είδους προγράμματα. Από 600 σε 800 είναι συμμετέχοντες τα τελευταία χρόνια. Και βλέπουμε επίσης ότι αν συγκρίνουμε με άλλες δομές, υπό το εθνικό δίκαιο ή όχι, πρόκειται για νομικά πρόσωπα, οπότε υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και μπορούν να αποφασίσουν εύκολα και να δράσουν γρήγορα. Με δύο λόγια, βλέπουμε ότι μπορούμε να αμβλύνουμε τις δυσκολίες από την διασυνοριακή διάσταση. Χρησιμοποιούμε αυτούς τους δείχτες, όπως είπαμε, και η εικόνα που παίρνουμε είναι πολύ θετική. Εμείς από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει ο ίδιος ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας. Ένα πράγμα ακόμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι τέλεια, γιατί εξακολουθούμε να βλέπουμε ότι χρειάζεται καλύτερη επικοινωνία. Πρόκειται για καινοτομία, για πολλές αρχές περιφερειακές και τοπικές Χρειάζεται λοιπόν περισσότερο συντονισμό μεταξύ των χωρών μελών για να τίθεται σε εφαρμογή ο κανονισμός και για να διασφαλίζεται ότι ο χειρισμός του ε, συνάδει με κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια. Αλλά αυτό είναι κάπως εκτός του κανονισμού. Έχει να κάνει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 ως ε, προηγούμενος ε, ε, γνωμοδότης, γνωμοδότης εισηγητής γνωμοδότης των ΕΟΕΣ πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο αποκτά, γίνεται όλο και πιο δημοφιλές. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ήδη 78 τέτοια οργαλεία και επίσης υπάρχουν διάφορα τα που συμμετέχουν σε αυτό. Βέβαια είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την διασυνοριακή συνεργασία και την περιφερειακή συνεργασία όπως ε, έχει προκύψει μέχρι στιγμής. Και αν υπάρξει λοιπόν μια ολοκληρωμένη γνωμοδότηση για αυτό, τότε αυτό το οποίο μας είπατε θα συνεισφέρει ακόμα πιο πολύ, ούτως ώστε το συγκεκριμένο εργαλείο να γίνει ακόμα πιο δημοφιλές και ακόμα πιο γνωστό και εν τέλει κάποιες ε, παρανοήσεις ε, οι οποίες ε, υπάρχουν σε διάφορες περιφέρειες για παράδειγμα στα ανατολικά σύνορα της Γερμανίας με την Πολωνία και την Τσεχία διότι εκεί υπάρχει ακόμα έλλειψη συνεννόησης, οπότε θα είναι καλό το να λυθούν αυτά τα προβλήματα και να χαιρετήσουμε αυτή την πρόταση. Ε, είδα και τον κατάλογο κριτηρίων της Επιτροπής και πιστεύω ότι θα τον εξετάσουμε λεπτομέρως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλα μέλη της Επιτροπής που θα θέλουν να κάνουν κάποιο σχόλιο. Όχι. Οπότε το ερώτημα είναι, υπάρχουν μέλη τα οποία θέλουν να ε, γύρουμε την ε, αντίρρησή μας πάνω σε αυτό ή μήπω να ζητήσουμε άλλου τρεις μήνε ε, για να σκεφτούμε τη συγκεκριμένη πρόταση. Όχι από ό,τι φαίνεται. Ε, πώς να καταλάβω αυτό που μου λέτε. Θέλετε επιπλέον χρόνο. Ωραία. Σημειώνουμε λοιπόν ότι θα πάρουμε λίγο χρόνο και κύριε Ζέλερ στην ε, περίοδο των τριών μήνων, ίσον και λιγότερο, το Δεκέμβριο μέσα, Το Δεκέμβριο λοιπόν θα το συμπεριλάβουμε στην ημερήσια διάταξή μας και αυτή τη φορά ελπίζω ότι η ε, πρόταση αυτή θα ολοκληρωθεί αυτή λοιπόν είναι η απόφασή μας σχετικά με, ε, το συγκεκριμένο κατεξουσιοδότη ε, κανονισμό και συνεχίζουμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάθεξης το οποίο αφορά την συζήτηση σχετικά με τι κοινέ διατάξει για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, συν το Ταμείο Συνεχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα και Αλληλείας και δημοσιονομικοί κανόνες για τα εν λόγω ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης κλπ. κλπ. Ο κανονισμό κοινών διατάξεων λοιπόν, CPR. Και σήμερα θα έχουμε την συζήτηση α, μετά την υποβολή ε, τροπολογιών που είναι γύρω στις 2.000 και παραπάνω. Η προθεσμία ήταν η 22 Οκτωβρίου. Η πρόταση αυτή είναι ίσως το πιο σημαντικό νομοθετικό κείμενο για την Επιτροπή μας και εξηγεί και το γιατί έχουν υποβληθεί τόσες πολλές τροπολογίες. Θα έχουμε επίσης τις ε, γνωμοδοτήσεις από 9, 9 συνολικά άλλες επιτροπές, οπότε ε, θα περιμένουμε ακόμα πιο πολλές τροπολογίες να λάβουμε. Σήμερα θα γίνει η συζήτηση στις κατατεθήσεις τροπολογίες και θα ακούσουμε επίσης την ε, θέση των εισηγητών διότι στη συνέχεια θα πρέπει να αποφασίσουμε για την ψηφοφορία σε αυτές τις νομοδοτήσεις, οπότε θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Κχέλ. Ο συνεισηγητής μου δεν είναι εδώ και εγώ περίμενα ότι θα ξεκινούσαμε αυτή τη συζήτηση λίγο πιο αργά. Όπως ε, είπατε, έχουμε 2.100 και κάτι τροπολογίες. Ε, τις διαβάζω ακόμα, δεν έχω τελειώσει τη μελέτη. Οπότε θα προτιμούσα να μην συζητήσουμε σήμερα για τροπολογίες. Παρ' όλα αυτά όμως ε, οι συνάδελφοι ήθελαν να μου δώσουν μια εικόνα. Αυτό το οποίο κατάφερα μέχρι στιγμής από τη γενική εικόνα ε, είναι ότι έχω να κάνω δύο-τρία σχόλια. Παρατηρώ λοιπόν ότι πολλές τροπολογίες θέλουν να προσθέσουν ε, στον ε, κανονισμό πολύ ωραία πράγματα, μεμονωμένα όλα είναι χρήσιμες, αξιόλογες ε, και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, όμως θεωρώ ότι αν θέλουμε απλοποίηση της πολιτικής συνοχής, της διοίκησης, της διαχείρισης, τότε δεν μπορώ να προσθέσω χιλιάδες πράγματα ακόμα. Παραδείγματα. Όταν ξεκινώ λοιπόν με τον ορισμό και λέω ότι θα πρέπει να έχουμε αυτές τις οριζόντιες αρχές ε, και να τα συμπεριλάβουμε και όλα και το ένα και το άλλο. Ναι, είναι χρήσιμο. Όταν όμω αναφέρω πολύ συγκεκριμένα πράγματα, αυτά τα πολύ συγκεκριμένα θα πρέπει να εξεταστούν και πολύ συγκεκριμένα. Οπότε θα πρέπει να γίνουν και άλλε ε, γνωμοδοτήσει ε, ως διοικού αρχή. Αυτό σημαίνει ότι ξαφνικά δημιουργώ ένα ολόκληρο κύμα ε, γραφειοκρατίας για να υποστηρίξω κάτι τέτοιο, όμως εν τέλει το αποτέλεσμα είναι ότι οι διοικητικές αρχές ε, ουσιαστικά τους δένουμε τα χέρια και χάνουμε κάθε ευελιξία που μπορεί να υπάρξει. Όταν παντού αναφέρουμε ότι ιδιαίτερο στις ε, βουνίσιε περιοχές, ε, τις ε, παράκτιες περιοχές θέλω να τις υποστηρίξω, τότε θα πρέπει όλο αυτό να το αποδείξω, διότι όταν το ζητάω τότε και η Επιτροπή θα πρέπει να συντάξει μια έκθεση σχετικά αν μπορεί να γίνει αυτό και με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουμε το αντίθετο από αυτό το οποίο ζητούσαμε, το οποίο είναι μια απλοποίηση και η ε, ευελιξία των περιφερειών. Επίσης, ε, δεν μπόρεσα να συνοηθώ ακόμα με τον κύριο Νόβακοβ. Η πρώτη μου αντίδραση λοιπόν ήταν ότι ε, στο πρώτο άρθρο απορρίπτω έτσι απλά όλες τις τροπολογίες διότι πολύ απλά σημαίνουν πολύ γραφειοκρατία. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη σημερινή ευκαιρία ούτως ώστε να κάνουμε στους συναδέλφους να καταλάβουν ότι δεν είμαι εναντίον κάτι από πολιτικής άποψης, αλλά επειδή θέλω να παραμείνει η ευελιξία στις περιφέρειες και αυτές να αποφασίζουν στο πλαίσιο μιας εταιρικής συμφωνίας, μιας ενισχυμένης εταιρικής αρχής, ε, μιας ε, στρατηγικής ανάπτυξης, ότι εκεί λοιπόν θα υπάρχει αυτό το οποίο πραγματικά θέλουν να κάνουν και ότι αυτό θα το διαπραγματεύονται με την Επιτροπή, θα ενημερώνονται γι' αυτό, όμως ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κι, άλλο, κι άλλη γραφειοκρατία γι' αυτό. Αυτό είναι το ένα σχόλιο και το άλλο είναι ένα βασικό πρόβλημα όπου θα πρέπει να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να έχουμε transfers ή όχι. Αύριο, όταν θα εξετάσουμε την γνωμοδότηση για το InvestEU και θα ψηφίσουμε για αυτό. Θα δούμε λοιπόν ε, πώς ε, στην Επιτροπή μας ε, είναι, πώς είναι η κατάσταση μεταξύ των δυνάμεων, αν μπορούμε να έχουμε κάποιον συμβιβασμό και τι κατεύθυνση μπορούμε να ακολουθήσουμε. Οπότε θα έλεγα ότι σήμερα δεν μπορούμε να το απαντήσουμε έτσι απλά αυτό. Επίσης όσον αφορά το άρθρο 15 ε, αυτό αφορά όλες τις κατευθύνσεις, όλες τις παρατάξεις. Ε, ε, έχουμε διαγραφή, έχουμε να προσθέσουμε κι άλλα, έχουμε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε είναι δύσκολο να βρούμε συμβιβασμούς πάνω σε αυτό. Οπότε και θα πρέπει να εξετάσουμε, να κάνουμε συζητήσεις. Έχουμε την πρώτη συνάντηση των σκιωδών για τις 4 Δεκεμβρίου, αν θυμάμαι καλά θα προσπαθήσουμε με συζητήσεις να βρούμε ε, μία οδό ούτως ώστε να διαπραγματευτούμε ε, συμβιβαστικές διότι το τελευταίο το οποίο χρειαζόμαστε είναι εν τέλει είναι ένα αποτέλεσμα μια ψηφοφορία στην Ολομέλεια όπου θα είμαστε διαχωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα οπότε καλό θα ήταν να έχουμε μια κοινή συζήτηση ούτως ώστε να ακολουθήσουμε μια κοινή ε, γραμμή γνωρίζοντας ότι γίνεται σε μια εποχή όπου ο καθένας ξεκινά την προεκλογική του εκστρατεία ε, και το οποίο έχει τις αντίστοιχες πιέσεις. Το τρίτο σχόλιο τώρα που θα ήθελα να κάνω είναι ότι πρόσεξα σε διάφορα σημεία ότι ε, ήδη έχει ασκηθεί πίεση έχει από κάποια κρατημέλη προς κάποιους ε, ευρωβουλευτές το οπότε περιμένω στους πρώτους τριμερείς διαλόγους ε, να φανεί αυτό οπότε θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι για να έχουμε ευελιξία στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο θα πρέπει να έχουμε μια θέση του Κοινοβουλίου Οπότε, πώς μπορώ εγώ να διαπραγματευτώ με το Συμβούλιο όταν το, τη θέση του Κοινοβουλίου ε, εμφανίζονται θέσεις του Συμβουλίου. Να πούμε ότι πώς θα μπορέσω εγώ να πω ότι πάμε σε αυτό, ότι μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμού σε κάποια σημεία και σε άλλα όχι. Όταν λοιπόν σε διάφορα σημεία ήδη ε, βλέπω ε, τη θέση του Συμβουλίου σε μένα, ε, τότε η διαπραγματεύσει θα είναι δύσκολος. Οπότε ελπίζω ότι η κατάσταση θα προχωρήσει έτσι, ούτω ώστε να μπορέσω να έχω ε, μια ευελιξία διαπραγματεύση. ακόμα και αν στο πίσω του μυαλού μου έχω ότι σε ένα βαθμό μπορούμε να μοιραστούμε κάποια θέση, σε κάποια άλλα σημεία όμως. Αυτό μπορεί να μην συμβαίνει. Και έτσι δεν θα μπορώ να διαπραγματευτώ. Δεν είμαι βέβαιη για όλες τις ε, τροπολογίες, αν ε, από νομική άποψη έχουν κάποιο νόημα, ε, οπότε αυτή τη στιγμή με τη Γραμματεία και με την Επιτροπή το ελέγχουμε για να δούμε τι μπορεί να γίνει και τι όχι, όμως αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να κάνω σχόλια για 2.000 τροπολογίες. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο μου σχόλιο σχετικά με τις τροπολογίες τις οποίες έχω λάβει. Για μένα όμως ένα είναι ξεκάθαρο ότι οι ε, περισσότερες τοπολογίες είναι τόσο μεγάλες και τόσο διαφορετικές που νομίζω ότι θα είναι αδύνατο το Δεκέμβριο να ψηφίσουμε για αυτές. Θα χρειαστούμε χρόνο ούτως ώστε να το συζητήσουμε αυτό με τους σκιώδες και πιστεύω ότι και οι παρατάξεις από μόνες τους χρειάζονται χρόνο διότι όπως είπα ε, σε ορισμένα σημεία υπάρχουν εντελώς αντιθέμενες απόψεις οπότε θα ήταν πιο λογικό να αφιερώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο ε, από ότι στο τέλος να βρεθούμε ε, σε ένα σκηνικό όπου η διαπραγματευτική θέση του Κοινοβουλίου θα είναι πολύ περιορισμένη. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μου ε, σχόλιο όσον αφορά τις τροπολογίες που μου δόθηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς ο συνεισηγητής δεν έχει φτάσει ακόμα, ίσως να εμφανιστεί αργότερα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους Σκιώδης να παρουσιάσουν τις δικές τους απόψεις μετά από την τοποθέτηση της κυρίας Κρέλ. Τόμασιτς δεν είναι εδώ. Θα ξεκινήσω εγώ ίδια ο Σκιώδης για τους φιλελευθέρους και θα μου επιτρέψετε να κάνω ορισμένα σχόλια. Να πω ότι πράγματι υποστηρίζω την ανάγκη που υπάρχει να υπάρξει άπλετος χρόνος για τη συζήτηση όλων των τροπολογιών και των πιθανών συμβιβαστικών. Δεν πιζόμεθα. Απαιτείται χρόνος για την αναζήτηση των σωστών λύσεων. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να μπορούσαμε να οργανώσουμε τις τροπολογίες και τα σχόλια επί των τροπολογιών σε ομάδες. Αυτό θα είχα κάνει για να προετοιμαστώ για τη σημερινή συνεδρίαση. Να πω ότι η πρώτη ομάδα των τροπολογιών που είχα προτείνει εγώ, νομίζω όμως κι άλλοι συνάδελφοι, ε, ζήτησαν το ίδιο πράγμα. Συνίσταται από τροπολογίες οι οποίες συνδέονται με περαιτέρω δεσμούς με το, Ευρωπαϊκ, με το ΦΕΟΓΑ το οποίο αυτή τη στιγμή δεν περιλαμβάνεται βέβαια στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορούμε να βρούμε έτσι λοιπόν τις συμβιβαστικές λύσεις ανάμεσα στους Κιώβης και τους συναδέλφους ε, οι οποίοι κατέθεσαν τροπολογίες. Οι υπόλοιπες τροπολογίες αφορούν τους στόχους για τις κλιματολογικές αλλαγές. Εγώ προτείνω το 30%. αντί για 25 το οποίο προτείνεται. Αυτή είναι η πρόταση την οποία κάνω και αυτό ακριβώς είναι και η βάση για τις συμβιβαστικές ε, λύσεις ανάμεσα στους κοιόδης. Οι υπόλοιπε ομάδες τοπολογιών δύσκολα θα συμβιβαστούν σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, διαφορετικές προτάσεις από εντελώς διαφορετικές πολιτικές ομάδες και είναι λίγο δύσκολο να υπάρξει κάποια συνεννόηση. Πάντως χρειάζεται χρόνος για περαιτέρω συζήτηση για να βρούμε μια κάποια ισορροπία δεν πρέπει αυτό το θέμα να μας οδηγήσει στην Ολομέλεια και να έχουμε διαιρεθεί πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σαν Ρέτζι σε μια λύση η οποία στο μέλλον να είναι αποδεκτή από την Ολομέλεια. Το ίδιο λοιπόν ισχύει σύνδεση και με τα υπόλοιπα μέσα και με τα χρηματοδοτικά μέσα είναι κάτι το οποίο έχει, εν πάση παρουσιάζει διαφορές. Ε, παρουσιάζουν διαφορές οι πολιτικές ομάδες και το ίδιο θα φανεί και στην Ολομέλεια. Εγώ είχα ως εισηγήτρια, ως σκιώδης εισηγήτρια προτείνει μία αύξηση των μεταφορών. Τώρα, σχετικά με τα επιμέρους, ε, επιμέρους χρηματοδοτικά μέσα, θα περιμένουμε τις ψηφοφορίες στη Ρέτζη για να δούμε ακριβώς ποια θα είναι η πλειοψηφία και θα δούμε ακριβώς τι θα, πώς θα εξελιχθούν οι προσπάθειες συμβιβασμού και για, το επόμενο, για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Αύξηση λοιπόν της προχρωματοδότησης, αύξηση των ποσών συνολικά για το Interreg. Ελπίζω να βρούμε κάποιες κοινέ λύσεις. Αυτή είναι η κατεύθυνση την οποία εγώ νομίζω ότι μπορούμε να επιδιώξουμε. Συμπερασματικά θα ήθελα να πω, όπως ακριβώς έχω ήδη πει, ότι έχω προτείνει αύξηση ε, των πιστώσεων και για τη διασυνοριακή συνεργασία, κοινή ονοματολογία και γενικότερα μέτρα τα οποία ευνοούν τους μεθοριακούς πληθυσμούς. Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία τίθενται και τα οποία νομίζω ότι δεν θα προκαλέσουν πάρα πολλές δυσκολίες. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το 25% συνιστά μία αρκετά περίπλοκη λύση. Λοιπόν, θέλουμε περισσότερο χρόνο, το υποστηρίζω αυτό και υποστηρίζω και την εισηγήτρια να προσπαθήσουμε να βρούμε μια συμβιβαστική πρόταση και κοινή απόφαση της Επιτροπής μας, όχι στην Ολομέλεια. Η επόμενη ομιλήτρια, Βάνα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και την ε, εισηγήτρια και φυσικά και τον συνεισηγητή ε, για την ε, δουλειά που γίνεται και για το γεγονός ότι σε πολλά σημεία στο προσχέδιο υπάρχουν πολλές από τις θέσεις της Επιτροπής μας. Ε, πιστεύω ότι θα υπάρξουν ε, συμφωνίες ούτως ώστε η αρχή της εταιρική σχέσης να ε, ενισχυθεί, το οποίο θέλουμε να φανεί και στο CPR, η ενίσχυση της προστασίας για το κλίμα, το οποίο αναφέρει και η Πρόεδρες, είναι κάτι το οποίο εμεί οι πράσινοι το θέλουμε περισσότερο και βλέπουμε ότι η συζήτηση πηγαίνει προ τη σωστή κατεύθυνση. Το άλλο σημαντικό για εμά και το γνωρίζετε ήδη από τι αρχικέ μα συζήτηση είναι οι οριζόντιες αρχές ε, να επανεισαχθούν και πάλι στον τομέα της ίσης μεταχείρισης ανδρών ε, και γυναικών στο πλαίσιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ε, βιώσιμων στόχων. Γνωρίζω ότι σε άλλους τους τομείς του CPR θα εμφανίζονταν αυτές οι αρχές και το βλέπουμε αυτό παρόλα αυτά ναι. όμως συγκεκριμένα όσον αφορά τα θεμέλια δικαιώματα, το κράτος δικαίου και όλα αυτά, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και αυτό. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό για την διασφάλιση της στήρισης αυτών των δικαιωμάτων να μην παρεκκλίνει ο ΣΥΠΙΑ από αυτό ε, το θέμα. Επίσης, ε, εκ μέρους της ε, παράταξής μου, δεν θα ήθελα να μιλήσω για τη δυνατότητα μεταφορών ε, σε άλλα εργαλεία, μακροοικονομικές προϋποθέσεις, το έχουμε συζητήσει. Το έχουμε συμπεριλάβει και σε άλλα πλαίσια και θα πρέπει όλα αυτά να τα συμπεριλάβουμε. Σήμερα θα ήθελα να αναφέρω ένα συγκεκριμένο σημείο ε, το οποίο, ε, για το οποίο θα ήθελα μια διευκρίνηση από την Επιτροπή το οποίο αφορά την σχέση με το ευρωπαϊκό εξάμεινο, το οποίο το βλέπουμε κάπως κριτικά και ιδιαίτερος όσον αφορά ε, ε, το, το, το, πλαίσιο ε, δεδομένων της Επιτροπής, το οποίο είδαμε τον Οκτώβριο και το οποίο βλέπει μια ενίσχυση των ευρωπαϊκών απαιτήσεων και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Βλέπουμε ότι μετά από αυτό το κατάλογο δεδομένων είμαι ιδιαίτερα ανήσυχη για αυτήν την κίνηση της Επιτροπής ε, διότι ιδιαιτέρως όσον αφορά τα οικονομικά και τα οικονομικά αυτά ε, θα αποφασίζουν, αυτός ο τομέας της Επιτροπής θα αποφασίζει ε, για τα κονδύλια που θα δίνονται στις περιφέρειες με αποτέλεσμα να αγνοούνται και να περιθωριοποιούνται ακόμα οι ανάγκες των περιφοριών ε, και φαίνεται ότι ε, και γι' αυτό το λόγο εμείς απαιτού, ε, απορρίπτουμε την συγκεκριμένη πρόταση της Επιτροπής. Εμείς θα θέλουμε περισσότερη διαφάνεια ε, και ιδιαιτέρως όσον αφορά, διευκρι... και ιδιαίτερου όσον αφορά τη συγκεκριμένη παρο... διαδικασία. Θα θέλαμε διευκρίνηση από την Επιτροπή σχετικά με το πώς θα εφαρμοστεί. Θα θέλαμε λοιπόν να ευχαριστούμε για τη συνεργασία και επίσης θέλουμε και εμείς συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ενισχυμένη θέση θέση της Επιτροπής είδα κάποιε τροπολογίες όπου τα κράτη-μέλη με τον έναν ή άλλο τρόπο προσπαθούν να περάσουν τα δικά τους ε, θέλω. Οπότε ε, πιστεύω ότι οι επιθυμίες των κρατών μελών ε, αντικατοπτρίζονται καλύτερα στο Συμβούλιο και εμείς θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Συνολικά λοιπόν συμφωνώ επίσης με το γεγονός ότι θέλουμε μια καλή βάση για διαπραγματεύσεις Χρειαζόμαστε χρόνο για αυτό, όμως δεν έχουμε πολύ χρονικό. Αν ε, έχω υπολογίσει καλά, η 14η Φεβρουαρίου θα είναι η τελευταία ε, προθεσμία που έχουμε για να το ψηφίσουμε και να προχωρήσει στη συνέχεια στην Ολομέλεια. Είναι λίγο ο χρόνο και γι' αυτό το λόγο επιθυμούμε ε, να δημιουργηθεί, να παρουσιαστεί ένα χρονοδιάγραμμα όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντεμάτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν είμαστε και πολύ εδώ, αλλά καλό είναι να ξεκινήσει η συζήτηση για τις τροπολογίες, που είναι πάρα πολλές. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι βλέποντας τις τροπολογίες των συναδέλφων, βλέπω να υπάρχει μια σύμπτωση στην βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στο Γεωργικό Ταμείο και τα υπόλοιπα διαφθορτικά. Πολλές φορές έχουμε ασκήσει κριτική στην επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ είχα προτείνει μια συνολική πολιτική για τα πέντε επενδυτικά αυτά ταμεία και οι προτάσεις ως έχουν στρεβλώνουν ουσιαστικά τους στόχους. Για τον μηχανισμό των transfers τώρα. Έχει προηγηθεί η διαβούλευση για το άρθρο 10 για την συνεργασία των διαρθρωτικών ταμείων με το InvestEU και περάσαμε από το 5 στο 2 με 3% και αυτό είναι κάτι το οποίο περιορίζει τις μεταφορές μεσοπρόθεσμα για το κίνημα των πέντε αστέρων και για το άρθρο 21 και για το InvestEU κάθε μορφή μεταφοράς των μέσων μας των οικονομικών ε, μπορεί να παραβιάσει την αρχή της εδαφικότητας. Οι πόροι οι οποίοι στρέφονται σε συγκεκριμένες περιοχές ή κατηγορίες περιοχών ε, και που γίνονται αντικείμενο διαχείρισης από άλλα μέσα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παραμείνει στην ίδια περιοχή. Δεν θα πρέπει τα ποσά να μετακινηθούν από τη μία περιοχή στην άλλη. Είναι δύσκολο να γίνει μια τέτοια μορφή μεταφοράς. Με τη ρήτρα εθνικής προστασίας ο μηχανισμός, ο ανταγωνιστικός στη συγκεκριμένη περίπτωση μεταφέρει από το ευρωπαϊκό επίπεδο στο εθνικό επίπεδο. Για χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία πολλές φορές έχουν εσωτερικές διαφορές μεταξύ τους πάρα πολύ μεγάλες. Για το άρθρο 15 τώρα, εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι και δεν έχουμε ξεκάθαρη άποψη για το θέμα της εμπλοκής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, ε, Εξαμήνου σε σχέση και με το άρθρο 15 και το 23. Δεν έχει αλλάξει η πρόταση σχετικά με την ισχύουσα πρόταση για τη την μακροερεσιμότητα σε σχέση με τα λειτουργικά προγράμματα στις περιφέρειες των χωρών που δεν σέβονται τις συστάσεις αναχώρα. Εμείς προσπαθήσαμε και με τις τροπολογίες μας να περιορίσουμε τις συνέπειες αυτές μέσω της τροπολογίας 49 σαν παράδειγμα που καθιστά υποχρεωμένη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώνει το Κοινοβούλιο, κάτι το οποίο θα ήταν καλό αλλά δεν είναι επαρκές. Και η δική μας τροπολογία διαγραφής του άρθρου 15 υπάρχουν συνάδελφοι πρασίνων, γκούε και σοσιαλιστών που έχουν τον ίδιο στόχο με τις δικές τους. Γι' αυτό παρακαλώ να σεβαστούμε την ψήφο της Ολομέλειας, της έκθεσης Βέστβαλ ε, της ε, Δευτέρα Ιουνίου του 2017, όπου είχαμε καταθέσει με τους πρασίνους πολλούς σοσιαλιστές και την Γκουε ε, μία τροπολογία απόρριψης της μακροαιρεσιμότητας, γιατί η Ρέτζη δεν είχε το θάρρος να το κάνει μόνη της. Κλείνοντας να πω ότι ο νέος κανονισμός θα πρέπει να δημιουργήσει και μια άλλη αιρεσιμότητα σχετικά με τις παραβάσεις γύρω από το άρθρο 91. Αυτή η αιρεσιμότητα είναι παρούσα στον προγραμματισμό 2010-2016 και 2016-2021, αλλά όχι στην παρούσα πρόταση. Μια μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναγνωρίζει ότι οι καταστάσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί δεν είχαν προβλεφθεί. Και γι' αυτό η τροπολογία μου 1766 ζητά να ληφθεί υπόψη η ερεσιμότητα ως αρνητικό χαρακτηριστικό. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα συζητήσουμε αναλυτικότερα βέβαια στον κατάλληλο χρόνο. Ευχαριστώ. Αυτά είναι τα σχόλια των σκιωδών. Θα δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Και εγώ νομίζω ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό έγγραφο αυτό το οποίο συζητάμε. Από τη μία είμαι ιδιαίτερος ευτυχής που ένας τόσο μεγάλος αριθμός τροπολογιών έχει κατατεθεί. Αυτό δείχνει ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά και θέλουν να, βελτιώσουν τον κανονισμό. Από την άλλη, μια τέτοια πολλαπλότητα προτάσεων ε, αποδεικνύει ότι κάποιες από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρκετά θεωρητικές και όχι τόσο πρακτικές. Εμείς θα θέλαμε να είναι καταρχάς βιώσιμες. όχι μόνο θεωρητικές προσπάθειες για τη μείωση των διαφορών ανάμεσα στις χώρες και τις περιοχές και υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, σε βάση περιπτώσει, στην πρόταση αυτή της Επιτροπής οι, όχι μόνο οι εθνικοί οργανισμοί αλλά και οι περιφέρειες θα πρέπει να εμπλέκονται στη διαχείριση των ποσών. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να έχουμε σημαντικές βελτιώσεις. Ξέρουμε ότι αλλάζουν βέβαια τα κόμματα στην εξουσία και οι κυβερνητικοί σχηματισμοί και κάθε νέα κυβέρνηση έχει νέες προτεραιότητες. Αν λοιπόν αποπειραθούμε να ορίσουμε με πιο συγκεκριμένο τρόπο το περιεχόμενο του κανονισμού, ίσως να πετύχουμε και καλύτερα τους στόχους μας. Ήδη από το 2016 έχουν επισυμβεί αρκετές διοικητικές αλλαγές σε πάρα πολλές χώρες και ιδιαίτερα στις περιοχές ΜΑΤ2 θα πρέπει ε, κάποιες αλλαγές να καλύψουν το σύνολο των χωρών. Δυστυχώς όμως λόγω των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι περιοχές του 2016 δεν θα υπάρχουν το 2027. Υπάρχει μια γεωγραφική ανακατανομή. Ε, οπότε και δεν υπάρχει αναφορά στις περιοχές αυτές ως έχει το κείμενο τώρα. Θα πρέπει να κατανοήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όλες οι αλλαγές που είχαν γίνει το 2018 θα πρέπει να γίνουν σεβαστές. Η δική μου χώρα, η Λιθουανία. Η χώρα μου διαιρείται σε δύο περιφέρειες και η διαφορά ανάμεσα στις δύο περιφέρειες αυτές είναι διπλού τύπου. Αν δεν δώσουμε λοιπόν την δυνατότητα για τη λιγότερο ευνοημένη περιοχή να αναπτύξει την οικονομία της, τότε οι διαφορές αυτές ε, μπορεί να μεγεθυνθούν το 2017. Εν πάση περιπτώσει, τυπικά οι στόχοι φαίνονται καλοί, αλλά αν δει κανείς πραγματικά τι συμβαίνει, η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική, γι' αυτό και θα καταθέσω προφορικές τροπολογίες. Θα ήθελα να τονίσω ότι ορισμένοι δεν κατανοούν κάποιες από τις προτάσεις. Σαν παράδειγμα, μια περιοχή η οποία καλύπτει τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους και ας συγκρίνουμε την περιοχή αυτή με μια άλλη περιφέρεια ε, στις οποίες οι δείκτες είναι χαμηλότεροι του μέσου όρου εκεί θα πρέπει σύμφωνα με τους κανόνες της προχρηματοδότησης ε, να υπάρξουν σημαντικότερες ε, επενδύσεις και προσπάθειες χρηματοδότησης. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει επιτέλους να πάρουμε κάποια απόφαση για το οποία θα είναι τα κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιούμε. Εφόσον όλα γίνονται επί τη βάση των περιφερειών, αυτό θα πρέπει να υπαγορεύει και τον τρόπο χρηματοδότησής τους. Αν πάλι επιθυμούμε να εξετάσουμε την κατάσταση με βάση τους εθνικούς μέσους όρους, ας το κάνουμε. Ίσως όμως έτσι κάποιες χώρες να μην είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν πλήρως τις υπάρχουσες δυνατότητες. Όταν λήξουν κάποια από τα προγράμματα χρηματοδότησης φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε πετύχει τη μείωση των διαφορών όπως τουλάχιστον θα το επιθυμούσαμε ανάμεσα στις περιφέρειες. Τα ποσά λοιπόν είναι αρκετά σημαντικά και ελπίζω να μπορέσουν να μειώσουν τις διαφορές ανάμεσα στις περιφέρειες αποφεύγοντας τις ε, μη χρειαζούμενες μορφές εσωτερικής μετανάστευσης. Κάποιοι εγκαταλείπουν, επαναλαμβάνω, τις περιοχές τους ε, λόγω ακριβώς της έλλειψης απασχόλησης. Το να υπάρχει λοιπόν σύνδεση ανάμεσα στα διαφορετικά ταμεία είναι κάτι πολύ σημαντικό και το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όλα αυτά θα πρέπει να, αν κάποιος θέλει να τα χρησιμοποιήσει, θα πρέπει να γνωρίζει καλά τους κανόνες, γιατί είναι διαφορετικοί οι κανόνες σε κάθε περίπτωση. Καλό θα ήταν να υπάρξει ουσιαστική εναρμόνιση ε, για όλα τα ταμεία των κανόνων. Σαν παράδειγμα, πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης, οι οποίες ξεκινούν από συγκεκριμένες τοπικές κοινότητες, οι πρωτοβουλίες αυτές λέμε ότι είναι εφικτές. Αλλά αυτή η διατύπωση δεν λέει και τίποτα. Όλα αυτά δεν θα εξαρτώνται, εν πάση περιπτώσει, από τις τοπικές αρχές, αλλά από τις κρατικές δομές οργάνωσης. Οπότε θα πρέπει να βελτιώσουμε λίγο τις δυνατότητες των περιφερειών. Και θα πρέπει ένα ποσοστό να στραφεί αποκλειστικά προς τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Έτσι με τον τρόπο αυτό όχι μόνο θα υπάρξει περισσότερη πρόοδος στη συνεργασία των περιοχών μεταξύ τους, αλλά θα αυξηθεί και τελικά το ποσό συνολικά που θα έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη. Αν λοιπόν πάνε καλά τα πράγματα σε περιφερειακό επίπεδο και αν διαχειριστούμε σωστά τις, τις περιφερειακές δυνατότητες, θα βελτιώσουμε και τους εθνικούς μέσους όρους. Αυτά τα ολίγα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι συνεισηγητές έχουν να αντιμετωπίσουν ένα περίπλοκο θέμα και σε πολύ περιορισμένο χρόνο. Δεν θέλω τώρα να παρουσιάσω τις τροπολογίες μου, αλλά να υπογραμμίσω τις τρεις προτεραιότητες τις οποίες προσπαθώ να προωθήσω μέσω των τροπολογιών μου. Η βασική προτεραιότητα, όπως και για άλλους συναδέλφους, έχει σαν στόχο την απλοποίηση της ζωής των δικαιούχων των διαχειριστικών αρχών είναι τροπολογίες τεχνικής φύσεως, οι οποίες όμως ε, μπορούν να πετύχουν πολύ συγκεκριμένες λύσεις και μάλιστα μία τροπολογία η οποία βοηθά το κόστος της επαλήθευσης των συνθήκων που ε, πρέπει να ευνοηθούν στις διάφορες περιοχές να μην αναλαμβάνεται από τους δικαιούχους και σε σχέση με τα χρηματοδοτικά μέσα και σε σχέση με την τεχνική βοήθεια. Μια δεύτερη προτεραιότητα αφορά την ίδια την αρχιτεκτονική και την μέθοδο κατανομής. Εδώ θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις προτάσεις τις οποίες έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σε μεταβατική φάση περιφέρειες. Η διεύρυνση η οποία προτείνεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία δεν είναι κάτι το αρνητικό αλλά θα ήθελα να επικαλεστώ την πρόταση των συναδέλφων να ευνοήσουμε το 70% σε επίπεδο προχρηματοδότησης. Και τέλος, είμαι διστακτικός σε σχέση με την πρόταση την οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο υπαλογισμού της περιφερειακής συνεργασίας, της εδαφικής συνεργασίας. Είδα μια εξομοίωση επί χάρτου. Είναι κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικότητες της εδαφικές και θα είναι κάτι το ιδιαίτερα αρνητικό όπου έχουν ιδιαίτερα υψηλή πυκνότητα πληθυσμιακή. Μια τελευταία προτεραιότητα είναι ότι μπορούμε μέσω των προτάσεων αυτών να στείλουμε ξεκάθαρα μηνύματα για το μέλλον σε δύο κυρίως θέματα. Πρώτον, σε σχέση με την κοινωνική Ευρώπη. Η κοινωνική Ευρώπη είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Καταθέτω τροπολογίες οι οποίες διασφαλίζουν ότι ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να τροφοδοτείται από συγκεκριμένα γεγονότα πραγματικά μέτρα για την καταπολέμηση της στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Και ένα άλλο θέμα το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε, είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα του Brexit. Όλες οι μελέτες τις οποίες έχουμε μέχρι σήμερα δείχνουν ότι ανεξαρτήτως της φύσεως των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ηνωμένου Βασιλείου, το Brexit θα έχει άμεσες συνέπειες στις περιφέρειές μας. Σε ορισμένες περιφέρειες, διότι θα καταστούν ουσιαστικά νέα σύνορα εξωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άμεσες συνέπειες και γενικότερα στις περιφέρειες οι οποίες έχουν συνδέσμους, εμπορικές σχέσεις με το Ηνωμένο, ε, με το Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ισπανία και στη Γαλλία. Εγώ ξέρω ότι πολλοί από τους συναδέλφους με τους οποίους συνεργάστηκα είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε σχέση με όλα αυτά. Τα είπαμε πολύ αναλυτικά και με τον Λάμπερτ. Ο ρόλος λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να είναι εδώ ουδέτερος. Πρέπει κατά κάποιο τρόπο το μήνυμα που θα στείλουμε να είναι ένα μήνυμα προστασίας και δεύτερον, η Ευρώπη έχει την δυνατότητα να προκαταλάβει και όχι να περιμένει να συμβεί κάτι. Μαζί με συναδέλφους λοιπόν κατέθεσα τροπολογίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα εξειδητευμένο ταμείο το οποίο θα στηρίξει τις περιφέρειες οι οποίες θα επηρεαστούν περισσότερο από το Brexit. Αυτά σύντομα σας τα είπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ επιμένω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ποιοτική προσέγγιση. Να έχουμε μια ισχυρή εντολή και γι' αυτό το λόγο καλό θα ήταν να αφιερώσουμε χρόνο ώστε να συζητήσουμε ε, λεπτομερέστερα όλες τις ε, τροπολογίες ε, διότι πραγματικά πιστεύω ότι θα έχει σημαντική επιρροή στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις οπότε καλό θα ήταν τώρα να αφιερώσουμε χρόνο και στη συνέχεια να μεταβούμε στην πρώτη ανάγνωση και να μην βιαστούμε. Ένα μόνο ερώτημα έχω όσον αφορά τις μεταφορές. Ναι, έχουμε πολιτικές διαφορές σχετικά με το αν συμφωνούμε στην εθελοντική φύση των μεταφορών ή όχι και ε, για το αν θα πρέπει να πάνε τα ποσά αυτά του Ταμείου Συνοχής ε, στο InvestEU. Όμως το ερώτημά μου προς τους συζητητές είναι έξυπνο το να ε, χάσουμε αυτή την δυνατότητα για να ενισχύσουμε τη θέση μας του τριμερείς ή θα ήταν ένα επιπλέον επιχείρημα για αυτές τις χώρες οι οποίες δεν θέλουν να αυξηθεί το κονδύλι και θέλουν ένα πιο μειωμένο κονδύλι για την ε, πολιτική συνοχής ή μπορούμε να πούμε ότι το Κοινοβούλιο δεν θέλει να μεταφέρει χρήματα ε, ε, στο Connecting Europe Facility και να πούμε ότι να έχουμε ένα άλλο επιχείρημα το οποίο θα ισχυροποιεί τη θέση μας. Αυτό είναι το ερώτημά μας. Λοιπόν, πώς μπορούμε να το ενσωματώσουμε αυτό στις συμβιβαστικές, διότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, λοιπόν, εν ώψη των τριμερών διαλόγων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ο κύριος Ποστινάρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. θα εφιστήσω την προσοχή σας ε, στο να αποτρέψουμε το χειρότερο σενάριο, δηλαδή την μεταφορά ε, όλων των υποχρεώσεων στο επόμενο κοινοβούλιο, το οποίο πραγματικά είναι το χειρότερο ε, σενάριο. Και σήμερα στην, στο Βουκουρέστι, ο κύριος Σταγιάννη κάλεσε την Ρωμανική Προεδρία να κάνει ό,τι μπορεί, ούτω ώστε να διασφαλίσει την πολιτική συμφωνία για το PΔΠ και να εγκριθεί ε, στη Σύνοδο του ΣΥΜΠΙΟ. Αυτό είναι η πολιτική συμφωνία. Ωραία και καλά. Αν όμως αφήσουμε όλους τους βασικούς κανονισμούς να περάσουν στο επόμενο κοινοβούλιο, τότε το νωρίτερο που μπορεί να γίνει αυτό θα είναι τέλη του 2021. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Εάν σε έξι μήνες, οι έξι μήνες δεν μας αρκούν για να αρχίσουμε να συζητούμε και να το ψηφίζουμε, τότε Πώς θα επιταχύνει τη διαδικασία το επόμενου κοινοβούλιο όταν, γνωρίζει ότι θα, όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια δραματική ανανέωση ε, του κοινοβούλιο το οποίο θα έχει διαφορετικά οράματα. Διακυβεύουμε λοιπόν το μέλλον της πολιτικής συνοχής αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας έστω μονάχα για την αγγλική εκδοχή, την αγγλογαλλική ούτως ώστε να αρχίσουμε να ψηφίσουμε οποιαδήποτε καθυστέρηση θα έχει σορευτικές συνέπειες το οποίο θα στοιχήσει στους πολίτες. Πολιτικά λοιπόν είναι ένα επικίνδυνο όπλο στα χέρια των ευρωσκεπτικιστών. Επίσης είναι σημαντικό όσον αφορά τις ερεσιμότητες και εγώ συμφωνώ με αυτούς που επανειλημμένως είπαν ότι θα πρέπει να αντιταχθούμε στις μακροαιρεσιμότητες γνωρίζοντας ε, την Ισπανική και την Πορτογαλική όθεση που αποτράπηκαν λόγω της δέσμευσης του Κοινοβουλίου. Για ποιο λόγο λοιπόν το Κοινοβούλιο να το ξανακάνει τη στιγμή που ξέρει ότι αυτό επηρεάζει μονάχα τους ανθρώπους και τις ε, περιφέρειες και όχι τις κυβερνήσεις. Τώρα, για το κράτος δικαίου τον κανονισμό για αυτό το θέμα. Ύστερα, από συζητήσεις με πολλούς συναδέλφους, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να βρούμε μια καλά σχεδιασμένη πρόταση. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, δεν θα επισέλθετε σε λεπτομέρειες, όμως να μην δίνει απεριόριστη δύναμη και εξουσία στην Επιτροπή. Αυτό είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει να απορριφθεί ε, αμέσως. Είναι σημαντικό αυτό για το Κοινοβούλιο και γι' αυτό το λόγο καλό το συνάδελφο Βαν Μίντελμπουργκ και όλους τους συναδέλφους ότι ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων θα επεξεργαστεί το συγκεκριμένο θέμα. Είναι σημαντικό λοιπόν να το συντάξουμε με τρόπο ούτως ώστε να εφαρμόζεται και να μην ε, επιβάλλει ε, σοβαρές κυρώσεις στις περιφέρειες και τους πολίτες. Τέλος, ωραία και καλά να τα σκεφτούμε όλα τα θετικά και να τα δούμε όλα ρόδινα. Όμως, ας επιστρέψουμε στην δήλωση της προηγούμενης εβδομάδας, στη συνάντηση μεταξύ Μέρκελ και Μακρόν. Είπαν το 2021 θα υπάρξει συμφωνία για τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Είμαστε τόσο αφελείς να πιστεύουμε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης δεν θα επηρεάσουν καθόλου ε, μέρη του ΠΔΠ. Εάν δεν απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα τώρα, αυτό το κοινοβούλιο, το οποίο έχει λάβει εντολή από τους πολίτες αρχίζουμε να ταξιδεύουμε σε αχαρτογράφητα ύδατα και διακυβεύουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, διότι η ε, πολιτική συνοχής αφορά την αλληλεγγύη. Με μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων δεν έχουμε τίποτα. Και δεν θα έχουμε μια, χωρίς μια ένα πλαίσιο για την πολιτική συνοχή, σαν ανοίγουμε το κουτί της, ε, της Πανδώρας. Αυτό λοιπόν είναι η παράκλησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να απαντήσω στο πρώτο σας σχόλιο και να σας πω ότι όταν μιλάμε για αρκετό χρόνο για συζητήσεις, δεν λέμε να ε, πάμε τις ψηφοφορίες για μετά τον Ιανουάριο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την δουλειά τους μέχρι στιγμής που είναι τρομερή η δουλειά που κάναν. Όμως θα ήθελα να πω ότι όλοι μας και οι σκιώδεις πιστεύουμε ότι η ψηφοφορία θα γίνει τον Ιανουάριο στην Επιτροπή. Οπότε δεν θα το αναβάλουμε. Σήμερα θα το αποφασίσουν οι συντονιστές να ολοκληρώσουν το χρονοδιάγραμμα για την ψηφοφορία στην ε, Ρέτζη και στη συνέχεια στην Ολομέλεια. Αυτή η απάντησή μου όσον αφορά το πρώτο σας ε, σχόλια και μαζί με τους ε, συνεισηγητές επικεντρωνόμαστε ούτως ώστε αυτό να γίνει έγκαιρα και να ολοκληρώσουμε το έργο πριν από τις εκλογές. Ο λόγος ε, τώρα στον κύριο Τόμασιτς ε, που είναι ένας από τους σκιώδεις. Η κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ πολύ, συγγνώμη που καθυστέρησα, όμως ήμουνα ε, σε μια άλλη επιτροπή. Και εγώ θα ήθελα να τονίσω τις τροπολογίες που αφορούν ε, τις ε, χώρες από την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Οι συγκεκριμένες χώρες βασίζονται στο, στην πολιτική συνοχή και οποιαδήποτε μείωση στη χρηματοδότηση και στη χρηματοδότηση ή χρηματοδοτικό κενό θα έχει αρνητικές συνέπειες στην οικονομία και κατά συνέπεια θα πρέπει να αντιδράσουμε εγκαίρως και αποτελεσματικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να αποφύγουμε αυτές τις αρνητικές συνέπειες. Πρώτον, η αύξηση ε, του ε, εθνικού ποσοστό χρηματοδότησης. Οι πιο αδύναμες περιοχές χρειαζόνται μεγαλύτερη όθηση για να μπορέσουν να φτάσουν τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές και αυτή είναι μία από τις προστιθέμενες αξίες και βασικές αρχές της πολιτικής συνοχής. Η αύξηση ε, του ποσοστού χρηματοδότησης από 15% στο 30% είναι μία από τις σημαντικότερες ανησυχίες μας και μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά εμπόδια στην εφαρμογή των ε, προγραμμάτων να δημιουργήσει επιπλέον άχθος για τις διοικητικές αρχές αλλά και τους υποφελούμενους. Δεύτερον, οι τα μειωμένα ποσοστά προχρηματοδότησης που πληρώνονται ετησίως ε, μειώνονται και φοβόμαστε ότι αυτό θα καθυστερήσει περαιτέρω την ομαλή ε, έναρξη της εφαρμογής. Ε, χρειαζόμαστε επιπλέον πόρους ούτως ώστε να, ενισχυθεί, να ενισχυθούν οι επενδύσεις για την πολιτική συνοχή και τρίτον οι κανόνες οι κανονές ε, που αφορούν το decommitment ε, θα επηρεάσουν την ε, απορρόφηση των πόρων, όμως συμφωνούμε ότι τα ποσά τα οποία αναφέρονται στο πι 21-27 θα βελτιώσουν την απόδοση και θα συνεισφέρουν σε μια αποτελεσματική διαχείριση και προστιθέμενη αξία. Και τέλος, το πι δέλτα πι είναι μια ευκαιρία να δείξουμε την δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών. Τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ούτως ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική ευημερία και η κοινωνική ευημερία όλων των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι αποτελεί προτεραιότητα. Με βάση το πολιτικό κλίμα και τι επερχόμενε εκλογέ θα πρέπει να δούμε, ε, ε, να έχουμε ένα ΠΔΠ το οποίο εξυπηρετεί τι κοινωνίε και βοηθά την ανάπτυξη. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υιοθέτηση του ΠΔΠ δεν θα έχει μόνο πολιτικές συνέπειες αλλά και πρακτικές διότι υπάρχουν πολλοί ε, που, ε, εποφελούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και θα έχουν ένα χρηματοδοτικό κενό και γι' αυτό το λόγο το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει πολιτική καθυστέρηση όταν θα ξεκινήσουν οι τριμεροί διάλογοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πόλτσακ τώρα. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θέλω να σας ε, ευχαριστήσω και να πω ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις, πιστεύω. Άκουσα αυτά που είπε και η προηγούμενη μιλήτρια. Πιστεύω πραγματικά ότι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση και ότι το τωρινό κοινοβούλιο που έχει μια συγκεκριμένη θητεία, όλοι μας έχουμε μια συγκεκριμένη θητεία εδώ, πρέπει να τελειώσουμε με αυτό το θέμα σε αυτήν τη θητεία. Τουλάχιστον εγώ αυτό στηρίζω. Ζούμε σε μια εποχή προκλήσεων απέναντι στην πολιτική συνοχής και δεν πρόκειται εδώ πέρα μόνο για το Brexit που θα έχει επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις, η κλιματική αλλαγή, τα κοινωνικά ζητήματα κλπ. Φυσικά μπορεί να ενδιαφέρουν οι απόψεις μας για το οι προκλήσεις αυτές τη θέση πρέπει να έχουν μέσα σε αυτή την πρόταση. Αλλά θα ήθελα το κείμενο σε πρώτη ανάγνωση να εγκριθεί στην δικιά μας ακόμα θητεία και εντολή. Ακούστηκαν διάφορες απόψεις σχετικά με την υπερβολική γραφειοκρατία όταν κινητοποιείται το Ταμείο. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια έχουν πάρει τελικά την ταμπέλα της υπερβολικής γραφειοκρατίας και για τους ε, δικαιούχους, ε, αυτούς τους οποίους προορίζεται η πολιτική αυτή, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Οπότε μέσα από αυτές τις τεχνικές τροπολογίες που πρότεινα, καμιά δεκαριά, θέλουμε την πολιτική αυτή συνοχής να την κάνουμε πιο φιλική για το χρήστη. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πάντως, αν ε, τα συγκρίνω με την γεωργική πολιτική. Εκεί η κατάσταση είναι πιο εύκολη, που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν το κείμενο αυτό να το προχωρήσουμε μέσα στην προθεσμία και κυρίως να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Νομίζω ότι είναι σωστό ο προσανατολισμό μα, αλλά μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Ο κύριο Φανβρέκα. Σωστά ή όχι. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Η κυρία Κρέλ πρώτα. Βέβαια, όποτε θέλετε. Έτσι, όπως πηγαίνει η κατάσταση, πιστεύω ότι συμφωνούμε ότι θα μπορέσουμε, να να έχουμε ένα αποτέλεσμα έγκαιρα. Ένα ερώτημα όμως ε, το οποίο ε, θα ήθελα να απαντήσω. Οι δύο συνεισηγητές πρότειναν στην Επιτροπή στο σχέδιο έκθεσης ότι δεν θέλουμε αυτές τις μεταφορές. Το είχαμε συμφωνήσει αυτό. Διότι αυτή θα είναι η maximum θέση ε, για την Επιτροπή, για τα κράτη-μέλη. Και στην αρχή είχαμε την εντύπωση ότι υπήρχε πλειοψηφία που το υποστηρίζει αυτό. Οπότε αύριο στην ψηφοφορία για το InvestEU θα δούμε ποιες είναι οι πλειοψηφίες ε, και στην Επιτροπή ε, θα πρέπει να προετοιμαστούμε για, κάποιες, για κάποιους συμβιβασμούς διότι όταν βλέπουμε τις τροπολογίες, ε, κάποιες έχουν γίνει δεκτές. Μερικές φορές ε, η επιθυμία είναι από διαπραγματευτικής άποψης να έχουμε καλύτερη θέση ούτως ώστε, ε, γιατί πλησιάζουν οι ευρωεκλογές. Επίσης πρέπει να τονίσω ένα πράγμα. έχω ένα βασικό πρόβλημα εγώ προσωπικά με, τα, με τις μεταφορές διότι αυτό αποτελεί παρέμβαση στην πολιτική συντοχής διότι μπορούμε να πούμε αυτό είναι καλό πρόγραμμα, το άλλο είναι καλό πρόγραμμα, οπότε παίρνουμε λεφτά από την πολιτική συνοχή. Αυτό δεν το τόλμησε ούτε η Επιτροπή, όμως ε, τώρα από την πίσω πόρτα βλέπουμε να εισάγεται θα μπορούσα να σας πω παραδείγματα όπου είμαι 100% βέβαιη ότι τα κράτη-μέλη περιμένουν να μπορέσουν ε, εθελοντικά να το χάσουν αυτό, διότι όταν το InvestEU δεν ε, πρέπει ε, να ε, λαμβάνει υπόψη του το κράτος μέλος, αλλά η πολιτική συνοχή στο κάνει αυτό, τότε ε, και υπάρχουν όλες αυτές οι αρχές ε, περί εταιρικής σχέσης και συμφωνίες, τότε υπάρχει πολύ πιο εύκολος δρόμος μέσω του Investigu για το κράτος μέλος. Και εδώ είναι που βλέπω τον κίνδυνο ότι από τη μία θέλουμε να οργανώσουμε μία σύγχρονη πολιτική συνοχή, η οποία δεν μπορεί να είναι η ίδια όπως πριν από 30 χρόνια, και από την άλλη πλευρά όμως θέλουμε πραγματικά να κάνουμε τις περιφέρειες να συμμετάσχουν και εδώ υπάρχει το πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο ήθελα μία ε, maximum θέση. Αύριο το αργότερο λοιπόν όμως με την ψηφοφορία θα δούμε ποιες είναι οι πλειοψηφίε και φυσικά στη συνέχεια και εγώ ε, θα πρέπει να ε, προσαρμόσω τις προσωπικές μου απόψεις ε, και σίγουρα εγώ με τον συνεισηγητή θα καταλήξουμε σε σε συμβιβαστικέ οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν το πώ είναι η εικόνα στο κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο αυτό δεν είναι όπως πριν από 7 χρόνια όπου συμφωνούσε ε, και ε, τσακωνόμασταν για κάθε ερασιμότητα και παρόλα αυτά χάναμε. Όμως θα πρέπει να δούμε τώρα τι έχει νόημα, τι είναι εφικτό, ποιο μα οδηγεί στη λάθο κατεύθυνση και εν τέλει πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε καλέ συμβιβαστικέ και θα λάβουμε την απαραίτητη πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ. Uh, yes. Ναι. Θα έδινα και σε εσά και στον κύριο Νοβακο το λόγο μετά από τον κύριο Φαρμπρέσκα. Αλλά έτσι κι αλλιώ θα σα ξαναδώσω το λόγο, εντάξει. Αν έχετε και θα έχετε σίγουρα κάτι να πείτε και μετά. Ο κύριο Φαρμπρέσκα τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ και τους δύο εισηγητές. Θα είμαι πολύ σύντομο, οπότε θα υπάρχει αρκετός χρόνος και για τους δύο, για να υπάρχει κι άλλος γύρος παρεμβάσεων. Και αυτό γιατί νομίζω ότι παρουσίασα την θέση μας και την προηγούμενη φορά εξήγησα πώς βλέπουμε εμείς τις δυσκολίες με τις τροπολογίες και γι' αυτό θα περιοριστώ σε τέσσερα ζητήματα τώρα. Το πρώτο, Θέλω να στηρίξω την κυρία Κρέλ που ζητάει απλοποίηση. Ξέρετε ότι η μεγαλύτερη κριτική της πολιτικής μας είναι ότι ακριβώς η πολιτική αυτή είναι υπερβολικά δύσκολη, γραφειοκρατική, επιβαρύνει υπερβολικά τους χρήστες. Και θα θυμόσαστε ότι προτείναμε 80 μέτρα απλοποίησης και από όσα άκουσα, τόσο από το Συμβούλιο όσο και από τις χώρες μέλη, τις διαχειριστικές αρχές κλπ, από ό,τι φαίνεται όλοι είναι θετικοί με αυτά τα μέτρα απλοποίησης. Για πρώτη φορά, είπανε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάει προς την σωστή κατεύθυνση, λιγότερος έλεγχος, λιγότερες επαληθεύσεις και περισσότερη ευελιξία για αυτούς που πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή τα μέτρα στην πράξη. 2.100 τροπολογίες. Καταλαβαίνετε και μόνο από το νούμερο αυτό καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Νομίζω ότι πολλές από αυτές τις τροπολογίες ακριβώς βοηθάνε να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία. Συνεπώς, σαφώς και στηρίζω την κυρία Κρέλ, την εισηγήτρια, στην έκκλησή της αυτή να είμαστε λογικοί και να επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτά που είναι σημαντικά για το σώμα και να περιορίσουμε όσο γίνεται αυτό που θα μας άρεσε μένουν να έχουμε, αλλά δεν είναι αναγκαίο ή περιπλέκει υπερβολικά τη ζωή των ανθρώπων που πρέπει να εφαρμόζουν την πολιτική στο μέλλον. Δεύτερον, κάτι που αναφέρατε αρκετοί από σας, τη σχέση ανάμεσα στα κονδύλια και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Μπορεί να μην είναι μεγάλη καινοτομία, αλλά πρόκειται για μια εξέλιξη που αλλάζει κάπως τα πράγματα σε σχέση με αυτό που προτείναμε. Βλέπουμε πολλές τροπολογίες οι οποίες ζητούν λιγότερες ή και καθόλου σχέση ανάμεσα στα κονδύλια και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Και εμείς πιστεύουμε ότι το αντίθετο χρειάζεται. Προσπάθησα και την προηγούμενη φορά να εξηγήσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα προσπαθεί να ξαναφτιάξει το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Δεν κοιτάει μόνο μεταρρυθμίσεις, κοιτάει και ανάγκες επενδύσεις, κενά σε επενδύσεις και εδώ τα κονδύλια αυτά έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Και θα στέλναμε ένα λάθος μήνυμα αν λέγαμε ότι η υπάρχουν οι διαδικασίες διακυβέρνησης στην Κεντρική Ευρώπη και υπάρχει η πολιτική συνοχής που δεν έχει καμία σχέση. Νομίζω ότι για το μέλλον της πολιτικής αυτό θα ήταν ένα μεγάλο στρατηγικό λάθος. Πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτό το εγχείρημα. Και ελπίζω να σας καθησυχάσω ε, λέγοντάς σας ότι δεν θα είναι η Γενική Διεύθυνση ΦΙΝ που θα έχει την διαχείριση. Έτσι καλώς, κανείς δεν θέλει να αλλάξει τα πράγματα. Αλλά έχει νόημα οι επενδύσεις μας να εξετάζονται στο γενικότερο πλαίσιο των δημοσίων επενδύσεων. Μιλάμε και για τις εθνικές επενδύσεις. Γι' αυτό αυτά τα δύο πρέπει να τα συνδέσουμε περισσότερο μεταξύ τους. Τρίτο, δεν συζητήθηκε τόσο πολύ εδώ σήμερα, αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικό για μας. Και έχει να κάνει με το πρώτο, δηλαδή είναι η ενδιάμεση αναθεώρηση. Υπάρχει μεγάλη ευελιξία στην πρότασή μας. Θα θυμόσαστε ότι οι αρχές μπορούν να αλλάξουν τις προτεραιότητες χρηματοδότησης χωρίς καν να πρέπει να περάσουν από την Κομισιόν για έγκριση. Άρα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και πιστεύουμε ότι έτσι καταλαβαίνει καλύτερο ο κόσμος τι συμβαίνει. Πιστεύουμε ότι έχει νόημα βέβαια κάποια στιγμή να καθίσουμε και να κάνουμε έναν απολογισμό και να αναθεωρήσουμε δεχομένω τα πράγματα εφόσον έχουν προκύψει νέε ανάγκε μετά από 7-10 χρόνια εφαρμογή. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό αυτή η αναθεώρηση στα μέσα του δρόμου να έχει πραγματικά νόημα, να είναι ουσιαστική και να μην ε, υπάρξουν ε, αλλαγές που να αμφισβητούν ε, την ίδια τη βάση και τα θεμέλια. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Είπαμε, Χρειάζεται σταθερότητα για τις επενδύσεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά έχει νόημα και σας υπενθυμίζω ότι η μεταναστευτική κρίση που δεν μπορούσαμε να βρούμε ούτε ένα ευρώ σχεδόν για να υπάρξει αναπρογραμματισμός, γιατί όλοι είχαν προγραμματιστεί στην Επιτροπή και τελείωσε. Αυτό για μας είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό η αναθεώρηση στα μέσα του δρόμου είναι πολύ σημαντική και θα στηρίξουμε τη θέση μας από αυτού. Τρίτο θέμα τώρα. Είναι η κάλυψη του CPR, του κανονισμού, γιατί εμείς τα χρήματα θα μπορούσαμε να τα πάρουμε από τη Γενική Διεύθυνση Home. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε όμως αυτό. Γιατί για άλλη μια φορά, εγώ δεν θέλω να μιλήσω για τους μηχανισμούς, αλλά αν έχετε μια μεταναστευτική κρίση, για παράδειγμα, έτσι, υπάρχει το θέμα της υποδοχής και της ένταξης των μεταναστών. Και εδώ είναι διαφορετικά τα κονδύλια. Είναι το κοινωνικό, είναι της περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά και της μετανάστευσης από τη Γενική Διεύθυνση Home. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα δούμε με συνοχή. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές. Αν κατάλαβα καλά από τις τροπολογίες, τώρα η δυνατότητα αυτή για το πρόγραμμα Invest EU επανέρχεται. Αντίθετα από ό,τι συνέβαινε πριν. Αλλά αν κατάλαβα καλά, η δυνατότητα αυτή διατίθεται μόνο από το 2025, μετά δηλαδή την ε, διάμεση αναθεώρηση. Για μας είναι αργά αυτό. Και δεν βλέπουμε γιατί να μην μπορούν οι χώρες μέλη, έτσι κι είναι σε θελοντική βάση, κανένας δεν είναι υποχρεωμένος. Γιατί να μην μπορούν λοιπόν να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτή την εναλλακτική νωρίτερα. Δεν θα αναφερθώ τώρα στις οικονομικές επιτυχίες, μόνο να υπενθυμίσω κάτι. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα στατιστικά δεδομένα, γιατί ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές που έχουν να κάνουν με την περιφερειακή ανάλυση, τα αίτια αναφοράς που χρησιμοποιούνται. Ό,τι έχουμε, έχουμε. Και δεν μπορούμε να τα αλλάζουμε υποθέτοντας ότι κάτι θα εγκριθεί αργότερα. Και να μιλάμε για εναλλακτικού τρόπους υπολογισμού της χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων, δηλαδή για τις χώρες μέλη. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω τώρα για τέτοια οικονομικά ζητήματα, γιατί είναι πέρα από το πεδίο που συζητάμε, τουλάχιστον το δικό μου. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Ωραία. Αυτά ήταν τα σχόλια. Α, ο κύριος Νόβαροφ πάλι μου ξέφυγε. Τον έχασα. Λοιπόν, εσείς κυρία Κρέλ τότε. Μια πρόταση μόνο παρακαλώ ακόμα όσον αφορά την μεταφορά στο Invest EU. Δεν αποφασίστηκε ακόμα, αλλά έχω την εντύπωση ότι καλύτερα είναι να σχεδιάσουμε ένα συμβασμό από το να μην έχουμε τίποτα. Καλύτερα συμβασμός παρά παραπάνω. Οπότε καλό είναι να το συζητήσουμε, αλλά δεν υπάρχει απόφαση ακόμα. Θα δούμε. Κατά τα άλλα, όπως είδατε, οι τροπολογίες μου θέλουν να χρησιμοποιήσουν κάθε δυνατότητα που υπάρχει ώστε το κράτος μέλος να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα στο Ταμείο Συνοχής και όχι η μεταφορά στο πρόγραμμα InvestEU. Αλλά όλα αυτά θα συζητηθούν στα πλαίσια κάποιου συμβιβασμού. Ίσως αύριο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριε Νοβάκοφ, θέλετε κάτι να προσθέσετε, όχι, όχι σε αυτό το στάδιο. Καλώς, μα μου λείψατε τόσο πολύ, περίμενα ότι θα έρθετε, θα πάρετε το λόγο και να, θα μας εξηγήσετε. Η κυρία Κρέλ το έκανε, εντάξει, ναι, ωραία, εντάξει. Δεν θέλετε, ωραία. Α, ναι, θέλετε. Ε, εντάξει, εγώ υπακούω στις εντολές τη Προέδρου. Θα πάρω το λόγο, δεν θα χάσω αυτή την ευκαιρία. Συγγνώμη που ήρθα τόσο αργά, αλλά καταλαβαίνετε είναι δύσκολη και στο Κοινοβούλιο αυτή την εποχή. Πολλές εκθέσεις, επιτροπές, ε, ψηφοφορίες, χρόνος, δύσκολο. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο κανονισμός κοινών διατάξεων είναι κάτι που θα μας απασχολήσει ακόμα ένα εξάμεινο. Και είναι ενδιαφέρον που τόσοι βουλευτές να ενδιαφέρονται. 2.100 τροπολογίε. 10 μέρες μου χρειάστηκαν για να διαβάσω τις τροπολογίε. Έχω υπόψη μου κάποιες ιδέες για συμβιβαστικές τροπολογίε, αλλά είναι κάτι που θα συζητήσω πρώτα με την κυρία Κρέλ, που είναι η συνεισηγήτρια. Και βέβαια και με τους σκιώδει συζητητές. Τώρα, και εδώ συμφωνώ με τον κύριο Ποστινάρο. Αυτή η διάθεση για καθυστέρηση είναι κάτι επικίνδυνο και χαίρομαι που η πρόεδρος μας μένει στην αρχική μας θέση, δηλαδή να ψηφίσουμε τον Ιανουάριο. Γιατί θα στέλναμε ένα λάθος πολιτικό μήνυμα, αν φαινόταν ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Και κανείς δεν θα δίνει σημασία στο Brexit ή οτιδήποτε άλλες δυσκολίες έχουμε. Αποτελέσματα θέλει ο κόσμος. Πιστεύω όμως ότι έχουμε αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε. Πάνε ήδη 6 μήνες που οριστήκαμε εισηγητές, οπότε προχωράμε. για τις μεταφορές των κονδυλίων. Θα είναι η καυτή πατάτα στη συζήτηση και δεν υπάρχει μια εύκολη απάντηση. Σίγουρα θα συμφωνήσετε όλοι και θα με στηρίξετε για το ότι κάπου πρέπει να βάλουμε ένα όριο για τις μεταφορές είχαμε όλοι πει ότι ήταν πολύ καλό πρόγραμμα η διευκόλυνση για την Ευρώπη, το συνδέοντα την Ευρώπη. Σύμφωνα, αλλά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα καλά προγράμματα. Το άερασμό για τους επιχειρηματίες, για παράδειγμα. Θα παίρνει χρήματα από τη συνοχή. Όχι, θέλουμε χωριστό προπολογισμό, χωριστή γραμμή στον προπολογισμό γι' αυτό. Πάντως το νιώθω, το βλέπω ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός στο μυαλό μου ποιος θα πάρει περισσότερο από το Ταμείο Συνοχής. Δεν ξέρω γιατί. Ήμασταν πολύ σκληροί για τη μεταφορά των 10 δισεκατομμυρίων στο συνδέοντα στην Ευρώπη και κάποιος είχε μια για 20. Περισσότερα. Φαντάζεστε, αν ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο, το συνολικό ποσό του Ταμείου Συνοχής θα είναι μικρότερο από ότι σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα αυτό θέλουμε, αυτό θέλει ο κόσμος, οι πολίτες. Μας κρίνουν όχι βάσει των λόγων μας, αλλά βάσει των πράξεών μας. Οπότε, ο κανονισμό αυτό κοινών διατάξεων και το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα αποδείξει πόσο πολύ πιστεύουμε στην Ευρώπη. Και αυτό ο ανταγωνισμό μεταξύ χωρών μελών, μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, είναι κάτι που δεν βοηθάει κανένα, παρά μόνο του λαϊκιστέ εκεί έξω. Πρόεδρο, ευχαριστούμε για όλη αυτή τη συζήτηση. Ναι. Θέλετε να μιλήσετε για την τροπολογία σας. Ναι, παρακαλώ. Ε, τι να κάνουμε, εδώ έχω κάνει μια πολιτική συζήτηση. Μα περί τίνο πρόκειται, τι είναι η περιφερειακή πολιτική, είναι να βάλουμε τα χρήματα σε ένα κουτί ή είναι θέμα επιδόσεων. Το Ταμείο Συνοχής δημιουργήθηκε για να επενδύσουμε σε υποδομές. Αν μπορούν να συνδυαστούν τα πράγματα, αν μπορούμε να πάρουμε χρήματα από το Ταμείο Συνοχής και να τα πάμε στην ε, διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, το ίδιο πράγμα λέμε. Για μένα το βασικό είναι στο τέλος, με όλους τους συμβασμούς που θα έχουμε, τελικά τι θα προσφέρουμε, πώς θα υποφεληθεί περισσότερο ο κόσμος, πού θα έχουμε την περισσότερη ευρωπαϊκή πρόσθετη αξία, πού θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για επενδύσεις. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το ποσό που συνδέεται με την πολιτική συνοχή σε αυτή καθ' αυτή ή με τις μεταφορές ή ο τσακωμός ανάμεσα σε επιτροπή, Εμένα με ενδιαφέρει να έχουμε αποτελέσματα και επιδόσεις. Να έχετε στο μυαλό σας ότι μερικές φορές έχουμε χαζούς τσακωμούς για το πώς να ονομάσουμε τα πράγματα, ενώ στην πράξη πρόκειται για προγράμματα. Ο κόσμος θέλει προγράμματα. Και αυτή είναι η γενική ιδέα των τροπολογιών τα επιπλέον 20 δις. Γιατί, γιατί όλοι οι πυρογνώμονε συμφωνούν, τουλάχιστον για την διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη, ότι προσφέρει αυτήν την προστιθέμενη αξία που όλοι τόσο χρειαζόμαστε στην Ευρώπη. Και αν δείτε το Ταμείο Συνοχής, δεν θα μας βοηθήσει στην Ευρώπη να έχουμε επενδύσεις για τους διαδρόμους. Πάλι θα επενδύσουμε σε εθνικά προγράμματα. Είμαι ευρωβουλευτής και προτιμάω να επενδύουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα και όχι σε καθαρά εθνικά προγράμματα. Το αστείο είναι ότι στην περίπτωσή σας και στη δικιά σας τη χώρα, η Βουλγαρία, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές. Οπότε θέλετε η Ευρώπη να βοηθήσει τη χώρα σα να επενδύσετε με την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη ή θέλετε να έρθουν οι Κινέζοι και να μπουν και να κάνουν αυτοί όλε τι επενδύσει. Εγώ προτιμάω την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Τώρα θα έχουμε την αντίδραση των συνεισηγητών. Πρώτα κυρία Κρέλ, μετά και ο κύριος Όλμπρεχτ έχει ζητήσει το λόγο. Ειλικρινά εκπλήσωμα. Αν εξετάσουμε το τι είναι το Ταμείο Συνοχής, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι δημιουργήθηκε ούτως ώστε να οργανώσει την Νομισματική Ένωση ε, και τις πιο ε, τις λιγότερο ανεπτυγμένες ε, χώρες να τις βοηθήσει ούτως ώστε να οργανωθούν με υποδομές περιβάλλον και ακριβώς για αυτόν τον λόγο επειδή αυτές οι χώρες έκαναν πρόοδους, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής μειώθηκε κατά 45%. Ε, όλο αυτό ε, δεν έχει να κάνει με ε, το, ε, η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη είναι κάτι υπέροχο, διότι ενώνει ε, την, ε, τις διάφορες περιφέρειες. Όμως θα πρέπει να ξέρετε ότι αρχής εξ αρχή υπήρχε ε, να ε, εξοπλιστούν τα διάφορα προγράμματα με τον απαραίτητο προπολογισμό, τον οποίο δεν θέλουν να χρηματοδοτήσουν τα κράτη-μέλη. Δεν θέλω να πω ποια είναι, αλλά όλοι γνωρίζουμε ε, ποια είναι. Η πολιτική συνοχής είναι κάτι διαφορετικό. Είναι συνδεδεμένη με τις συνθήκες και πρέπει να οργανώνει ούτως ώστε οι περιφέρειες οικονομικά, κοινωνικά και περιφερειακά να μπορέσουν μεταξύ τους να εξισορροπηθούν. Είναι μια διαφορετική προστιθέμενη, ε, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Είναι διαφορετική, αλλά έχει και αυτό ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Όμω δεν θα πρέπει να κάνουμε το λάθος να υπολογίσουμε, να αξιολογούμε το ένα ει βάρο του άλλου. Το δύσκολο αυτή τη στιγμή είναι ότι θα πρέπει να τα βγάλουμε πέρα τώρα με λιγότερα χρήματα και περισσότερες υποχρεώσεις από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Εάν είχαμε τα χρήματα έτσι όπως τα ήθελε το Κοινοβούλιο, τότε δεν θα χρειαζόταν να συζητούμε, να συζητούμε για τέτοια θέματα. Θα είχαμε και τα δύο προγράμματα, και το CEF, ε, και το Horizon ε, και πολλά πολλά άλλα και την πολιτική συνοχή, θα τα είχαμε όλα και δεν θα είχαμε το πρόβλημα λοιπόν ότι όλα θα πρέπει να τσακώνονται ε, για έναν προϋπολογισμό ο οποίος δεν φτάνει σε κανέναν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν το λύνουμε όταν εμεί κατηγορούμε ο ένα τον άλλον λέγοντα εσύ δεν κάνει αρκετά για την Ευρώπη και εσύ δεν κάνει αρκετά για την Ευρώπη. Και νομίζω ότι ω Επιτροπή εμεί έχουμε την ευθύνη μα απέναντι στην πολιτική συνοχή και παρεπιπτόντω η Βουλγαρία φυσικά ω μία από τι χώρε όπου όλε οι περιφέρειες δεν είναι τόσο ανεπτυγμένε ε, μπορεί να, χρειαστεί, ε, μπορεί να εκμεταλλευτεί τα χρήματα και να τα χρησιμοποιήσει τόσο από το Ταμείο Συνοχής όσο και από το CEF και για ποιο λόγο ε, η Βουλγαρία να δώσει χρήματα στο CEF. Και επίσης η σημαντικότερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ε, προκύπτει όταν καλύπτουμε ε, τα χάσματα μεταξύ των κρατών μελών και τα οποία δεν θα λυθούν αποκλειστικά και μόνο με το CEF. Διότι οι, οι διοικητικές αρχές πολλές φορές δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ετοιμότητα των κρατών μελών και να οργανωθεί έτσι ούτω ώστε ε, αυτά τα διασυνοριακά εμπόδια που υπάρχουν ε, να επιληθούν. Και αυτό λοιπόν δεν είναι ζήτημα χρημάτων. Μπορώ να θυμηθώ ένα πρόγραμμα μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας το οποίο πάγωσε για χρόνια και το πρόβλημα δεν ήταν η έλλειψη χρημάτων για τον οποίο δεν προχώρησε. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι όπου ένας κατηγορεί τον άλλον, εσύ είσαι καλύτερος, εγώ είμαι καλύτερος ή εγώ σκέφτομαι τις καλύτερε ιδέε, Δεν λειτουργεί έτσι, οπότε θα πρέπει να ε, σκεφτόμαστε λιγάκι πιο ενσωματωμένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ είναι και για μένα ε, δύσκολο να ε, λειτουργώ ως ε, πρόεδρος, διότι είμαι και σκιώδης και αναφέρθηκε επανειλημμένο στη Βουλγαρία. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σπάνιο να αναφέρεται η Βουλγαρία τόσο πολλές φορές. Θα ήθελα λοιπόν να προσθέσω κάτι στο ερώτημα του κυρίου Βαν Μίλτεμπουργκ. Όταν μιλάμε για την Βουλγαρία και τις επενδύσεις ε, στις υποδομές της Βουλγαρίας όπου υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη για την χώρα, για την ανάπτυξη της χώρας. Η Βουλγαρία όμως είναι μικρή χώρα στο μέσο των Βαλκανίων και η δραστηριότητα με τους γείτονές μας είναι το βασικότερο ερώτημα για την ανάπτυξη της Βουλγαρίας. Οπότε ίσως μία από τις πιθανές λύσεις θα ήταν ναι, το CEF. Όμως για διασυνοριακά προγράμματα τα οποία θα επιτρέψουν κάποιες μικρές, ε, μικρομεσαίες ε, χώρες όπως η Βουλγαρία να επενδύσουν χρήματα από το Ταμείο Συνοχής ε, και για αναπτυξιακά προγράμματα με τους γείτονες Βλέπω λοιπόν την δυνατότητα συμβασμού χρησιμοποιώντας και το παράδειγμα της Βουλγαρίας. Κύριε Ολμπρέχτ, ζητήσατε τον λόγο. Παρακαλώ. Λατρεύω αυτή τη συζήτηση, διότι επιστρέφουμε στην... στα βασικά. Οπότε θα ήθελα να πω κάτι αρχικά. Αν ακολουθήσουμε τη γραμμή του ε, Ματίας ότι μιλάμε για, το, για την πολιτική συνοχή. Ισχύει όλες οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ αφορούν τη συνοχή. Για τη συνοχή της Ευρώπη δεν χρειάζεσαι καθόλου πολιτική συνοχή και γι' αυτό το λόγο η Ολλανδική κυβέρνηση δεν θέλει να έχει ε, πολιτική συνοχή. Συνάντησα την πρέσβυρά σα και μου είπε ότι οι κατοχώρε δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την πολιτική συνοχή. Γιατί? Διότι αυτό είναι το εργαλείο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιούμε για τους αδύναμους. Όμως αυτό το οποίο τοπικές κυβερνήσεις ή καλύτερα οι τοπικές αρχές στην Ολλανδία γνωρίζουν ότι τα χρήματα αυτά λειτουργούν υπό τη μορφή της μόχλευσης και προς, κατά κάποιο τρόπο προσελκύουν περαιτέρω επενδύσεις. Τώρα για, τις, ε, ε, για το Ταμείο Συνοχής ήμουν δήμαρχος και έπαιρνα μέρος και στο Συμβούλιο των ε, Δήμων και Κοινοτήτων που συζητούσε τα του Μάστριχτ. Το Ταμείο Συνοχής βέβαια δημιουργήθηκε ειδικά για να βοηθήσει τις ασθενέστερες χώρες να προετοιμαστούν για την Ευρωζώνη να έχουν μεγάλες επενδύσεις, να μειώσουν γενικά την καθυστέρησή τους. Και αυτό ε, ίσχυε για χώρες οι οποίες ήταν κάτω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό του ευρωπαϊκού ΑΕΠ η cohesion policy. Κάτω από το 90%. Το θέμα λοιπόν είναι η μέθοδος την οποία αυτή τη στιγμή ε, μας απασχολεί, έτσι όπως είπε και η Κόνσταντς ε, Σκρέλ. Το θέμα είναι να υπάρξει σωστή ε, κατάρτιση, σωστός προγραμματισμός. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά συνοχή. Όλα αυτά μπορούν να ελέγχονται από τις Βρυξέλλες φυσικά. Υπάρχει η δυνατότητα να τα συγκεντρώσουμε όλα σε, επίμονο, σε επίπεδο διαχείρισης, ναι. Αλλά το αποτέλεσμα όμως ε, δεν είναι δεδομένο ότι θα επιτευχθεί. Έχουμε να κάνουμε με κάτι το διαφορετικό. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε κάποιες λύσεις σε τοπικό επίπεδο. Και όταν ο Επίτροπος Κάλλας είχε προτείνει να πάρουμε χρήματα από τη συνοχή και να την μεταφέρουμε στο ΣΕΦ το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί ειδικά για διαμεθοριακές και ψηφιακές συνεργασίες. Ο Βικτόρ Μποστινάρου ήταν τότε εισηγητής και μας είπε ο κύριος Κάλλας ότι το έκανε για προσωρινό λόγο αυτό και δεν θα το ξαναέκανε, δεν θα χρειαζόταν να το ξανακάνει. Γιατί? Γιατί υπήρχαν κάποιες συγκυρίες που το απαιτούσαν προσωρινά. Το ερώτημα λοιπόν σήμερα είναι το εξής. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν έβαλε από την αρχή τα χρήματα που έπρεπε στη συγκεκριμένη περίπτωση και γιατί δεν το ε, ενέταξε στον εθνικό, αν θέλετε, στο εθνικό κομμάτι χρηματοδότησης. Αυτό είναι λάθος. Όταν παίρνει κανείς χρήματα από τη συνοχή και το βάζει κάπου αλλού, τότε περνάει από τη μία πολιτική στην άλλη, από τη μία δε μέθοδο στην άλλη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαν να το κάνουν από πριν και να το πετύχουν από πριν. γιατί στην αρχή προτείνουν να το βάλουν στο συνολικό εθνικό ποσό και μετά να το βγάλουν από το ποσό αυτό ε, εκνευρίζοντας ιδιαίτερα τις κυβερνήσεις. Λοιπόν, γι' αυτό νομίζω ότι η ιδέα γενικά δεν είναι σωστή. Το Περιφερειακό Ταμείο είναι λίγο διαφορετικό. Ας προσπαθήσουμε να δούμε λοιπόν πώς θα καταστρέψουμε την πολιτική συνοχή. Άμα παίρνουμε από τη συνοχή και τα βάλουμε στη γεωργία, τα βάζουμε στην έρευνα, τότε όλα θα τα αποφασίζουν οι Βρυξέλλες, όλα θα τα κάνουν οι Βρυξέλλες. Μπορεί να τα κάνουν και πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα, αλλά θα καταστρέψουμε την περιφερειακή πολιτική. Νομίζω ότι το Περιφερειακό Ταμείο είναι ένα ταμείο κοινή διαχείρισης, από κοινού διαχείρισης. Αυτή είναι η λογική. Οπότε δεν έχει νόημα τα χρήματα αυτά να περνούν στο ΣΕΦ. Θα τα αυτά τα χρήματα από την συνοχή. Νομίζω λοιπόν ότι η ιδέα είναι, ακούγεται ωραία, αλλά έχω και άλλες ιδέες από πού μπορούν να έρθουν τα χρήματα αυτά. Ας τα πάρουμε από τα ΣΕΦ λοιπόν και να τα βάλουμε στο Περιφερειακό Ταμείο, γιατί όχι. Και αυτή η ιδέα είναι πολύ δημιουργική, όπως και η προηγούμενη. Ας σταματήσουμε λοιπόν να λέμε τα ίδια και τα ίδια. αλλά μιλάμε στα πλαίσια της ε, Ρέτζη και η Ρέτζη είναι υπέρ της αποκοινού διαχείρισης. Αυτή είναι η λογική μας, αυτή είναι η πολιτική μας. Δεν θέλουμε εμείς να φύγουμε από την πολιτική συνοχή, γιατί τότε τι θα μείνει από την πολιτική συνοχή. Ας κλείσουμε την πόρτα και σκοθούμε να πάμε όλοι σπίτια μας. Ευχαριστώ κύριο Πρόεδρε. Είναι καλό να, σας, να ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει άλλες ε, επιτροπές, στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού για παράδειγμα, έχουμε μία ενημέρωση σχετικά με το πώς τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν μέσα στο που προβλέπονται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής ε, για την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών ε, δικτύων μεταφορών. Το έκαναν λοιπόν με βάση των ε, μεταφορών από τα κράτη-μέλη. Όμως, εν τέλει έχτισαν το εσωτερικό δίκτυο και εκεί που θα έπρεπε να είχαν, ε, να είχαν υπάρξει ε, διασυνοριακές ε, γραμμές 15 με 20 χιλιόμετρα πριν από τις σύνορα σταματούσαν τις, τα έργα. Αυτό δεν είναι ευρωπαϊκή σκέψη. Είναι προγράμματα τα οποία, για τα οποία γίνονται σχεδιασμοί εδώ και 20 χρόνια Ωραία, καλό να χρησιμοποιηθούν ε, στο εσωτερικό που μπορεί να αποφελήσει κάποια επιχείρηση συνδρομικών γραμμών, όμως θέλουμε συνδέσεις ασχέτως του πώς είναι τα σύνορα, θέλουμε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να μπορούν να πηγαίνουν από τη μία χώρα στην άλλη γρήγορα. Και γι' αυτό το λόγο σας προειδοποιώ τα μέσα του Ταμείου Συνοχής να τα διασπάσουμε σε μεμονωμένα μικρότερα ε, μέσα, τα οποία εν τέλει θα υποφελούν μόνο τα κράτη-μέλη και εν τέλει να μην βοηθούν καθόλου στην συνοχή, στην ευρωπαϊκή συνοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε κύριο Ευχαριστώ. Μου είχε λείψει αυτή η συζήτηση. Είναι πολύ καλό που είχαμε αυτή τη συζήτηση. Είναι μια από τι καλύτερε που έχουμε κάνει σε αυτή την Επιτροπή. Πολύ τη χάρηκα, πραγματικά. Κάποια παρέμβαση τη Πρόεδρου εκτό μικροφώνου. Κρίμα που έχασα το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, λέει ο κ. Νοβακό. Αναφέρθηκε πολλέ φορέ η Βουλγαρία. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Μόνο ο κ. Σόλμπρεχτ δεν αναφέρθηκε στην Βουλγαρία, αλλά την ξέρει καλά. Ο κύριος Φαν Μίλτεμπορκ είπε ότι είναι υπέρ της Ευρώπης. Άρα υπέρ της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Τσεχίας κτλ. Που είναι πολύ καλό. Πολύ καλό να ξεκινάμε έτσι τη συζήτηση. Και αφού είναι υπέρ της Ευρώπης, καταλαβαίνει ότι η θεωρία των ε, εκείνων ε, των δικαιούχων που έχουν καθαρά κέρδη αυτών που είναι καθαροί εισφορείς είναι μια παλιωμοδίτικη συζήτηση. Τώρα για τον κύριο που μιλάει για μεταφορές από το Κοινωνικό Ταμείο στην διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη ή από το Ταμείο Ανάπτυξης της Υπέθρου ή και από το Ταμείο Λίας. Ναι, αλλά αυτό δεν τελειώνει πουθενά. Ποτέ. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε την οτροπία του ανταγωνισμού προς αυτή την κατεύθυνση και να αναγνωρίσουμε ότι αν σταματήσει η πολιτική συνοχής, σταματάει και ο τρόπος με τον οποίο σωματώνει τις διάφορες χώρες μέλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να ξέρετε, οι Κινέζοι θα λύσουν τα προβλήματά μας αν εμείς σταματήσουμε να χρηματοδοτούμε από το Ταμείο Συνοχής. Και καταλαβαίνετε γιατί. Ποτέ δεν είναι απλά τα πράγματα. 70% των πάντων που επενδύονται από το Ταμείο Συνοχής πήγαινε πίσω εκεί από όπου προήλθε ο κονδύλι. Αλλά σίγουρα θα καταλήξουμε σε κάποιον ισορροπημένο συμβιβασμό. Με πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πολύ. Πολύ χάρηκα αυτή τη συζήτηση. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πράγματι πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση και σίγουρα και οι συν ε, την εκτίμησαν πολύ. Ήταν η πρώτη ε, συζήτηση. Περιμένουμε τις συμβαστικές τροπολογίες και θα χρησιμοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι τον Ιανουάριο με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν το τελευταίο θέμα που είχαμε στην ημερήσια διάταξη για σήμερα. Αύριο το πρωί θα συνεχίσουμε στις 9. Τώρα έχουμε συνεδρίαση συντονιστών που θα αρχίσει σε 15 λεπτά. Στις 6 παρατέταρτο. Ή να ξεκινήσουμε τώρα. Μπορούμε τώρα, είναι εδώ συντονιστές. Μπορούν οι συντονιστές. Συμφωνείτε. Α, ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε περνάμε στη συνεδρίαση των συντονιστών και παρακαλώ τους προσκεκλημένους μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οποιοδήποτε σχόλιο συμμετέχει στη συνεδρίαση των συντονιστών να βγει από την αίθουσα παρακαλώ.